Κυρίες και κύριοι, μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Να ξέρετε ότι το σημείο 9 που έχει να κάνει με τον Τελωνιακό Κώδικα της Ένωσης, καθώς επίσης και με τα εμπορεύματα τα οποία έχουν εγκαταλείψει προσωρινά τα ταλουνιακά δάφη της Ένωσης, διαθαλάσσιας αέρος, έχει αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση. Το ίδιο ισχύει και για το σημείο 16, το οποίο είναι η συζήτηση για τις κανονιστικές, νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσει προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Αυτά τα δύο σημεία λοιπόν αναβάλλονται για τον Νοέμβριο, σωστά. Ωραία, οπότε με την διαφορά αυτή μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Ωραία. Και έτσι έχει ελαφρύνει κάπως η ημερήσια διάταξη για σήμερα το απόγευμα. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι ε, υπάρχει web streaming, δηλαδή μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίασή μας, ότι το newsletter είναι διαθέσιμο και εξετάζει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή της νομοθεσίας που έχει να κάνει με την προστασία των καταναλωτών. Πολύ σημαντικό. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε την ε, ένατη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας μας αύριο για την ε, ενιαία αγορά. Ιδιαίτερα, μάλιστα, θα κοιτάξουμε τις νέες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το roaming και για τα telecom, τηλεπικοινωνίες και δικαιώματα των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Θέματα που έχουν να κάνουν με τα ωφέλη, τις ευθύνες των καταναλωτών σίγουρα θα συζητηθούν. Οπότε αύριο το πρωί να έρθετε παρακαλώ 9.30. Α, όχι, όχι, την Τετάρτη διορθώνει ο Πρόεδρος. Την Τετάρτη το πρωί είναι αυτό. Θέλω να καλωσορίσω εδώ την κυρία Μπέρτε, η οποία αντικαθιστά τον, τον Κόρκας, που θα μου λείψει, γιατί δουλεύει τόσο σκληρά, λοιπόν και εσείς θα πρέπει να δουλέψετε τουλάχιστον εξίσου σκληρά. Κάθριν, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και προσβλέπουμε στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τώρα. Πρακτικά. Αν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αυτής δεν έχουν υπάρξει ενστάσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Και ένα άλλο θέμα, ενημέρωση για τριμερείς διαλόγους, δεν υπάρχει τίποτα. Σωστά. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία. Έχει καλώς. Ωραία. Έτσι είναι απλά τα πράγματα, γιατί φτάνουμε έτσι αμέσως στο σημείο 6, το οποίο αναφέρεται σε ένα πρόγραμμα της Ένωσης, προκειμένου να υποστηριχθούν συγκεκριμένες δραστηριότητε με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στην ε, χάραξη ενωσιακή πολιτικής στον τομέα τη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την περιοδο 2010 2017-2020. Βάσει του άρθρου 54, η ΕΚΟΝ βέβαια είναι αρμόδια, αλλά με αποκλειστική αρμοδιότητα για θέματα δημοσιονομικά και επιμερισμένες αρμοδιότητες για τα άρθρα 1 που έχει να κάνει με το θέμα και το πεδίο εφαρμογή, το 2 που έχει να κάνει με του στόχου και το 3 που έχει να κάνει με τους δικαιούχους. Αποκινούμε την ΙΜΚΟ λοιπόν, την Επιτροπή μα, εφόσον πρόκειται για θέματα σχετικά με του καταναλωτέ. Επί μακρό εγώ και ο κύριο Γκαλτιέρη που είναι ο πρόεδρος της ΕΚΟΝ συζητήσαμε για τι αρμοδιότητε. και καταλήξαμε στη συμφωνία ότι η τελική ψηφοφορία για δημοσιονομικά ζητήματα θα πρέπει να βρέχεται μετά από συνένεση μεταξύ των δύο επιτροπών. Ενδιαφέρον. Κανένας δεν ε, ε, ήθελε να γράψει σχετική έκθεση, οπότε η πρόεδρος το κάνει. Τώρα, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας να συνεχίσει να αντικατοπτρίζει τις ε, επιθυμίες και τις ανησυχίες των πολιτών. Κυρίως όταν πρόκειται για νομοθεσία που επηρεάζει τους καταναλωτές, είναι πάρα πολύ σημαντικό η δικιά μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή να εμπλέκεται. Γιατί αλλιώς θα διαπιστώσουμε κάποια στιγμή ότι κανείς δεν μας ακούει και συνεπώς οι καταναλωτές θα διαπιστώσουν ότι δική τους η φωνή δεν ακούγεται. Πρέπει επίσης να ελέγχουμε το έργο της ΕΚΟΝ, ότι βγαίνει δηλαδή από την Οικονομική Επιτροπή. Για το συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με χρήματα από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προκειμένου να πληρωθούν δύο οργανώσεις των καταναλωτών η Finance ε, Watch είναι η μία. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχουν τα χρήματα αυτά προκειμένου οι δύο αυτές οργανώσεις να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Η Finance Watch και η Better Finance είναι οι δύο οργανώσεις. Και είναι σημαντικό. Πρέπει οι καταναλωτές να έχουν φωνή, να ακούγονται. Όμως έχω κάποιες ανησυχίες γιατί έτσι όπως έχει διατύπωση τώρα λέει ότι μόνο οι δύο αυτές οργανώσεις μπορούν να υποφεληθούν από τη χρηματοδότηση. Και εγώ θα ήθελα να παραμείνει πιο ανοιχτό το θέμα. Να μπορούν και άλλες οργανώσεις ενδεχομένω να ζητήσουν χρηματοδότηση από αυτό το κονδύλιο. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές θα επωφεληθούν όσο γίνεται καλύτερα από τα χρήματα τα οποία απευθύνονται σε αυτούς και στις οργανώσεις τους και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Κλείστε τα κινητά σας, λέει η Πρόεδρος. Το άρθρο 2 λέει ότι οργανώσεις καταναλωτών πρέπει να είναι σε θέση να εκπροσωπούν τους καταναλωτές, αλλά δεν είναι σαφές από τη διατύπωση του κανονισμού πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό. Για παράδειγμα, προτείνω να συνδέονται με τα δίκτυα καταναλωτών που υπάρχουν ανά την Ευρώπη, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εκπροσωπούν τους καταναλωτές. Και ότι επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι καταναλωτές επίσης θα μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε διαβούλευση λαμβάνει η χώρα. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της και τρίτα μέρη, γιατί έχουν υπάρξει και ενστάσεις από τρίτες πλευρές μέσω των οργανώσεων αυτών, οπότε είναι σημαντικό να συμμετέχουν και τρίτα μέρη. Επίσης πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία. Οι δύο αυτές οργανώσεις σχολιάζουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εκείνη η οποία θέτει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι δύο αυτές οργανώσεις μπορούν να σχολιάσουν. Ε, αυτό για μένα δεν είναι καλό, υπάρχει κάποια αντίφαση εδώ. Πρέπει να υπάρχει αρκετός βαθμός ανεξαρτησίας για το έργο των οργανώσεων που χρηματοδοτούνται. Επίσης θα ήθελα και μία ρήτρα αναθεώρησης που να προσθεθεί στο άρθρο 9. Ένα άλλο ζήτημα δεν έχει να κάνει με αυτές τις οργανώσεις τόσο, αλλά με άλλες ομάδες στις Βρυξέλλες, που κανονικά συγχρηματοδοτούνται. Ο κανονισμός λέει ότι 60% της χρηματοδότησης θα έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τα υπόλοιπα από αλλού. Εγώ θα έλεγα το υπόλοιπο να μην έρχεται από κάποιο άλλο ευρωπαϊκό οργανισμό, γιατί τελικά θα είναι μόνο χρήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είτε απευθεία είτε μέσω οργανισμών που χρηματοδοτούνται από αυτήν, θα πηγαίνουν τα χρήματα στις οργανώσεις. Οπότε εγώ θα έλεγα να λέει ότι να υπάρχει συσσωρευτικά 60% χρηματοδότηση είτε έμεσα είτε άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή μπορούμε να βάλουμε αν θέλετε το έμεσα με κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό. Αλλά πάντως η χρηματοδότηση υπόλοιπη να γίνεται από μια τρίτη πλευρά, να μην γίνεται πάλι μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι λοιπόν τα κύρια σημεία που είχα να πω. Κατά τα άλλα, ελπίζω να συναντηθώ με τον εισηγητή της ΕΚΟΝ. Ξέρω όμως ότι υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις μέσα στην ΕΚΟΝ. Από το ΕΛΚ η Εύα Πάνοβα. Ε? Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ εγώ την κυρία Βαϊντέιρα που είναι σκιώδης εισηγήτρια. Όταν συμφώνησα με αυτό, η φωνή μου ήταν κάπως καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα, οπότε λυπάμαι που θα δείχω κάθε τόσο. Συγγνώμη. Λοιπόν, Πρώτον, το ΕΛΚ στηρίζει απόλυτα το στόχο της πρότασης αυτής. Πράγματι, είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα και να φροντίσουμε αντίστοιχα να διαμορφώνουμε τις πολιτικές μας. Και αυτό φυσικά πρέπει να γίνει με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Η σκέδωση συζήτητα θέλει να επιστήσει την προσοχή σας σε κάποια σημεία σε κάποια σημεία βλέπει περιθώριο βελτίωσης. Το πρώτο, δεν είναι πεπισμένη ότι δεν υπάρχει λόγος να αφισβητήσουμε ότι δύο αυτές οργανώσεις, η Better Finance και η Finance Watch, που πρέπει να είναι δικαιούχοι, κάνουν καλή δουλειά. Όμως, δεν είναι πεπισμένη ότι είναι ανάγκη να αναφέρονται τα ονόματα των δύο αυτών οργανώσεων μέσα στο κείμενο. Αυτό το νομοθετικό προτείνει να επικεντρωθούμε στους στόχους και στις απαιτήσεις για τους δικαιούχους. Η κυρία Βεντέιρα επίσης έχει και κάποιες επιφυλάξεις για το σημείο 3 του άρθρου 3 και για τους δύο δικαιούχους και τις λειτουργικές συνέπειες. Πολλοί νομίζω, συνάδελφοι, συμφωνούν ότι προκειμένου να βελτιωθούν οι οικονομικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό να ακουστεί περισσότερο η φωνή των καταναλωτών και άλλων τελικών χρηστών καθ' όλα τα στάδια της διαδικασίας. Γι' αυτό και πιστεύει ότι όσον αφορά τις δραστηριότητε των δικαιούχων θα ήταν καλό να έχουμε μια μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Ίσως με πιο στενή συνεργασία ε, με τους καταναλωτές από ανατολικές ε, χώρες, χώρες κεντρικής Ευρώπης ή τις βαλτικές χώρες. Θα ήταν σημαντικό για να ενισχυθεί ο ρόλος των τελικών χρηστών και των καταναλωτών. Και τέλος, έχει και κάποιες ανησυχίες για τη συγχρηματοδότηση των δικαιούχων. Όπως υπόθηκε, και δύο αυτές οργανώσεις εξαρτώνται πάρα πολύ από την κοινωτική χρηματοδότηση. Θα ήθελε λοιπόν να ακούσει περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Και τέλος, η σκιώδης εισηγητριά μας προσβλέπει σε καλή συνεργασία και με τον εισηγητή και με τους άλλους σκιώδες εισηγητές για να καταλήξουν όλοι μαζί σε πιο συγκεκριμένες προτάσεις προς εφαρμογή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ναι. Για τεκμέρους κυρία Μπολτζάνα, κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ. Να ξέρετε ότι έχει κάποια σχόλια που θα ήθελα να ακουστούν εδώ από τους συναδέλφους. Οι δύο οργανώσεις εδώ, η Finance Wars και η Better Finance, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική, για τους καταναλωτές, για τους αποταμιευτές, για τους επενδυτές και βοηθούν να γίνει περισσότερο κατανοητή η ευρωπαϊκή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή πολιτική. Δεδομένης της οικονομικής κρίσης, αν λάβουμε υπόψη μας ε, το έργο τους, καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί ένα καλό αντίβαρο στο οικονομικό λόμπι που πολλές φορές έχουμε εδώ. Και οι δύο αυτές οργανώσεις έχουν ένα τεράστιο δίκτυο με συμμετέχοντες και επίση έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές και για τους τελικούς χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το έργο τους το κάνουν πολύ καλά και αιτήσεις εκθέσεις τους είναι θετικέ. Οπότε οι σοσιαλιστές συμφωνούν με την πρόσωπα Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την δημοσιονομική ευθύνη και για τους πόρους που παρέχονται. Ευχαριστώ πολύ και θα στηρίξουμε την πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καθήν Ευχαριστώ. Μόλις ε, έφτασα και σας ζητώ συγγνώμη αλλά ε, η συνάδελφος δεν μπορεί να είναι εδώ, οπότε την αντικαθιστώ. Συμφωνεί απόλυτα, μας είπατε και εσείς, Πρόεδρε, για τους περιορισμούς σχετικά με τη χρηματοδότηση κτλ. Αλλά πριν ε, να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί αυτού. Πιστεύει ότι πρέπει να τονίσουμε ένα στοιχείο πολύ ξεκάθαρα. Αυτό το ταμείο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέσο να χρησιμοποιηθεί για πολιτικές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά του εμπορίου, κατά της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή, ε, στην ε, Finance Watch ε, ανοίχουν πάρα πολλές αριστερές οργανώσεις και συνδέονται τα ονόματά τους πολύ στενά με τις δράσεις κατά της TTIP. Έτσι λοιπόν, ενώ θέλει να υποστηρίξει την υπεράσπιση και την προστασία των καταναλωτών απέναντι στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, δεν θέλει ε, φυσικά να καταστήλει την ελευθερία της έκφρασης και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί δράσεις πέρα από το πεδίο εφαρμογή. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να το αποσαφηνίσουμε αυτό στους κανονισμούς και η Κομισιόν θα πρέπει να εγγυηθεί ότι γίνεται σεβαστή αυτή η αρχή όταν θα εγκρίνει το ετήσιο προγραμματισμό και για τις διοργανώσεις κάθε οργάνωση πρέπει να θυμόμαστε ότι θα λάβει ως ε, ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο και αυτό δεν θα πρέπει να είναι λευκή επιταγή για τις οργανώσεις αυτές. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο για αυτό το θέμα. Η Κομισιόν, μήπως θα ήθελε το λόγο για το ζήτημα αυτό, παρακαλώ. Πρόσωπος της Κομισιόν, ναι, ευχαριστώ. Λέγομαι Λιβεσέλες από την Γαμαδελτά Φίσμα. Είμαι υπεύθυνο ε, για αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστούμε που η Επιτροπή έχει την ευκαιρία να το συζητήσει αυτό το θέμα σήμερα. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια απλή και ξεκάθαρη πρόταση, γιατί ουσιαστικά συνεχίζει κάποια πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσεις ε, που είχαμε τα προηγούμενα πέντε χρόνια πριν να καταθέσουμε νέα πρόταση προκειμένου να χορηγήσουμε μια πιο σταθερή χρηματοδότηση σε αυτές τις δύο οργανώσεις. Θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχει η πίεση του χρόνου. Θα πρέπει να λάβουν αυτές οι δύο οργανώσεις χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ήδη στην αρχή του επόμενου έτους. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει δύο επιτροπές να γνωμοδοτήσουν επί της πρότασης αυτής, αλλά θα σας ευγνωμονούσα αν θα μπορούσατε να επιτυχύνετε τις εργασίες σας, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να είναι και σε θέση να εθετήσει την τελική του γνωμοδότηση κοντά στην ημερομηνία της έγκρισης του προπολογισμού του 2017, καθώς η πρόταση αυτή εν μέρη συνδέεται με τον ίδιο τον προπολογισμό σας. Ευχαριστώ. Um, Πρόεδρος, πώς θα μπορούσατε να απαντήσετε τις ερωτήσεις που ακούστηκαν από τους βουλευτές, ιδίω το θέμα που τέθηκε σε σχέση με το ότι θα διασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια θα δαπανηθούν ε, για την παροχή συμβουλών για θέματα καταναλωτή. Εγώ κατανοώ ότι στην νομοθεσία μας λέμε το θέμα ότι δίνουμε συμβουλές για καταναλωτικά ζητήματα και ουσιαστικά να δούμε και τι γίνεται ε, στην οδηγία προσπέκτους. Έχουμε από την ΠΕΟΚ πάρα πολύ ε, μεγάλη η δυνατότητα παροχή συμβουλών, αλλά όχι από αυτές τις δύο οργανώσεις. Μήπως θα μπορούσατε να αναφερθείτε λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα. Υπήρχε μια ερώτηση λοιπόν προς την Κομισιόν. I had a very opposite experience because I got very... Κοιτάξτε, εγώ έχω τις ε, αντίθετες πληροφορίες όταν ε, εργαζόμουν με ανάλογη νομοθεσία στην ΕΚΟΝ. Απλώς ε, ήθελα να αναφέρω ότι ήταν πολύ διαφορετική δική μου εμπειρία γιατί κάποια στιγμή δεκτήκαμε λόμπι και πώς λάβουμε αυτές τις πληροφορίες, το πώ λαμβάνουμε αυτέ τις πληροφορίες, ειδικά για του καταναλωτέ, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πώ λοιπόν μπορούμε να το διαχειριστούμε για να ασφαλίσουμε ότι ενίοτε ε, ουσιαστικά είναι καλέ οι πληροφορίε ε, και άλλε φορέ, ουσιαστικά έχουμε και κάποιε οργανώσει καταναλωτών που θα μπορούσαν να αναλάβουν το ίδιο έργο. Κοιτάξτε, και οι δύο συναδέλφοι αναφέρθηκαν στο πώς θα χρησιμοποιούνται τα κονδύλια ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ να απαντήσω τις ερωτήσεις σας, αν και έχασα την πρώτη, γιατί άργησα λίγο και ζητώ συγγνώμη. Πράγματι πιστεύω σε ό,τι αφορά τον στόχο της καθολικής πολιτικής. Τώρα κατανοούμε ότι αυτές οι δύο οργανώσεις ε, συνεισφέρουν ε, προκειμένου στο να υπάρχει μια πιο ισορροπημένη φωνή στην διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν αληθεύει ότι εξέδωσαν πάρα πολλές γνωμοδοτήσεις και έγγραφα για διάφορα νομοθετήματα, κυρίως ε, στο πλαίσιο της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όμως, επειδή είναι περιορισμένοι οι πόροι, οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν την ε, δυνατότητα να γνωμοδοτούν για όλα τα νομοθετήματα και ιδίω για τα νομοθετήματα που προέρχονται από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ και είναι και πολύ άριθμα τα τελευταία έτη και σε κάποιο βαθμό συμφώνησαν πάνω κάτω να γίνει κατανομή του άκθους ε, μεταξύ της Bacon και της Better Finance και της Finance Watch, έτσι ώστε να εξηγήσουμε ότι η BOIC ουσιαστικά θα ήταν περισσότερο αρμόδια για την πρόταση προσπέκτους. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δαπάνηση, το πώς θα δαπανηθούν τα κορδίλια, η Κομισιόν έχει θεσπίσει ένα κλασικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή η νομοθετική πρόταση θα παρουσιάζει την καθολική δομή, κυρίως σε ό,τι αφορά το στόχο και τα καθήκοντα αυτών των δύο οργανώσεων και η Κομισιόν ως κύρια αρμόδια αρχή εκτέλεσης του προπολογισμού θα λειτουργήσει και το πρόγραμμα. Αλλά όπως λέμε και στο άρθρο 5, αυτό θα γίνει βάση του προγράμματο εργασία που θα πρέπει να καταθέτουν ετησίω οι δύο και θα αξιολογείται από την Κομισιόν προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι σέβεται τους καθολικού στόχους ε, αυτών των δύο οργανώσεων. Επομένως, συνειδητοποιούμε το ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι θα σεβαστούμε το στόχο και τα καθήκοντα, όπως ε, αναγράφονται στα άρθρα και 2. Τα τελευταία πέντε χρόνια έτσι έχει συμβεί, γιατί πριν προχωρήσουμε στις τελικές πληρωμές, αξιολογούμε την έκθεση δραστηριότητας. Και ουσιαστικά αυτό το σε εξωτερική μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρσι και γνωμοδότησε αρκετά θετικά για τα καθήκοντα αυτών των οργανώσεων και για τις επιδόσεις τους. Και τέλος, προτείνουμε χρηματοδότηση για τα έτη 2017-2020, συνολικό ποσό κοντά στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα δαπανηθεί ετησίως και θα διαιρεθεί μεταξύ των δύο οργανώσεων. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο θα λαμβάνουν λίγο λιγότερα χρήματα και μόνο το 60% της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι μάλλον χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το 60%, το 40% θα πρέπει να το φροντίσουν οι ίδιες οι οργανώσεις, αλλά τουλάχιστον ε, θα πρέπει να έχουμε κάποια ξεκάθαρα στοιχεία για το ότι για τέσσερα χρόνια θα έχουν ε, χρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ζητήσουν και άλλους χρηματοδότες να προσθέσω κάτι. Εγώ όταν ε, εργάστηκα ε, στην Προσπέκτους ε, κάποιος εργαζόταν από αυτή και κάποιος άλλος. Γι' αυτό λέτε ότι δεν είναι να έχουμε το χάρη διαφορετικές οργανώσεις. Και θα ήθελα να αναφερθώ και στην ερώτηση από το ΕΛΚ. Θα πρέπει να αναφέρουμε το όνομα αυτών των οργανώσεων ή θα πρέπει να αφήσουμε ανοιχτό αυτό το θέμα έτσι ώστε να μπορούσε να συμμετάσχει και κάποια άλλη οργάνωση σε αυτό το πρόγραμμα. Και επίσης αναφερθήκατε στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίω. Και ξέρω, έχουμε κάποια χρόνια υψηλότερο ποσό, κάποια χρόνια χαμηλότερο. Μήπω ε, θα πρέπει να δούμε και αυτό το θέμα τη ευελιξία. Έχετε κάποιο σχόλιο σε σχέση με το αν θα πρέπει να αναφέρουμε το όνομα των οργανώσεων αυτών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Πολύ σκόπιμη η ερώτησή σα. Ε, την συζητήσαμε μακρόν με του ε, νομικού εμπειρογνώμονε και του δημοσιονομικού εμπειρογνώμονε. Το συμπέρασμα ήταν ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να τι κατονομάσουμε. Επίση, ε, βασιζόμαστε κυρίως στο ιστορικό των πέντε τελευταίων ετών. Γι' αυτό αποφασίσαμε να προτείνουμε στο Σύμβουλο και στο Κοινοβούλιο να χορηγήσουμε χρηματοδότηση απευθείας σε αυτές τις διοργανώσεις, γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια κάθε φορά οργανώναμε ένα διαγωνισμό και δεν υπήρχε κανένας άλλος υποψήφιος. Έτσι λοιπόν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ίσως να μην υπάρχουν τέτοια συγκρίσιμα κέντρα εμπειρογνωμοσύνης. Βέβαια αυτό μετά το 2020 δεν σημαίνει ότι θα ισχύει το ίδιο, αλλά για τα επόμενα τέσσερα χρόνια προτείνουμε την άμεση χορήγηση χρηματοδότηση σε αυτές τις δύο οργανώσεις και εγώ δεν πιστεύω ότι βέβαια είναι απαραίτητο να τις κατονομάσουμε στον ίδιο τον κανονισμό. Και καθώς αναφερθήκατε και στα χρήματα που θα δαπανούνται κατά χρόνο, τα ποσά που αναφέρονται στην νομοθετική πρόταση είναι τα ανώτατα όρια Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να εκτεμιεύσουμε και να χορηγήσουμε αυτό το ποσό κάθε χρόνο μέχρι το νοτοτόριο. Αυτό θα εξαρτάται από την αξιολόγηση του προγράμματος εργασίας και της ε, έκθεσης αξιολόγησης της ετήσιας έκθεσης αξιολόγησης δραστηριοτήτων. Ίσως ε, λοιπόν η τελική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι και μικρότερη από αυτή που αναμέναμε. Δηλαδή καταβάλουμε τα κονδύλια μόνο αν γίνει σωστή δουλειά. Και έχει φυσικά και υλοποιηθεί. Ελπίζω να απάντησα. Πρόεδρος, επομένως το χρονοδιάγραμμα θα είναι στενό. Γιατί θα ε, πρέπει ουσιαστικά να λάβουμε υπόψη και την ψηφορία στην ΕΚΟΝ ε, και στο Κοινοβούλιο και τον Δημοσιονομικό Κύπλο. Ε, στις ε, στις Οκτωβρίου έχουμε την προθεσμία και η προθεσμία για τροπολογίες 10 Νοεμβρίου, αλλά μόνο στα αγγλικά. Αλλά μόνο... Έτσι λοιπόν, επειδή είναι τόσο στενά τα χρονικά όρια, αν κάποιος έχει προτάσεις που θα ήθελε να τις εξετάσω εγώ, όταν θα συντάξω το πρώτο σχέδιο έκθεσης, θα μου τα στείλετε με email. Και ίσως να υπάρχουν βέβαια κάποιες διαφορετικές απόψεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα που συζητήθηκαν εδώ, αλλά ευχαρίστω να προσπαθήσω να συμπεριλάβω στο δυνατόν περισσότερα σχόλια και στον πρώτο γύρο. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της σημερινής διάταξης. το οποίο είναι η έκθεση Εύα Πάνοβα για το ε, Ευρωπαϊ... για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Υπολογιστικό Νέφος. Ε, ο κύριος ε, Σαφχάουσερ είναι ο εισηγητής της Ήτρε και έχει αναστείλει την ψηφοφορία έτσι ώστε η ΙΜΚΟ να μπορεί να συνεισφέρει, να έχει χρόνο. Αυτή η γνωμοδότηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σκόπιμη καθώς θα έχουμε μία νομοθετική πρόταση της Κομισιόν για την ελεύθερη ε, κυκλοφορία των δεδομένων. Και πράγματι αυτή η πρωτοβουλία για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων με τον κύριο Τίνκερ ε, είχαμε ουσιαστικά ένα ετήσιο διάλογο και είπε ότι ο κύριος ε, Επίτροπος αυτή είναι η κύρια προτεραιότητά του για το επόμενο έτος. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην Εύα Πάουνοβα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω το σχέδιο αυτό. Κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό και για τους ερευνητές, τους επιστήμονες, τη δημόσια δίκηση και γενικά για τους ε, πολίτες και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι από εσά, αλλά να τα ξαναπώ ίσως, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα απ' όλα τίμασε κάτι πριν από καιρό σχετικά με το ηλεκτρονικό νέφος προκειμένου να είμαστε σίγουροι ότι οι επιστήμονες, οι πολίτες μπορούν να υποφεληθούν από την επανάσταση αυτή κατά κάποιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως υπήρχαν κάποια εμπόδια τα οποία μας εμπόδιζαν να υποφεληθούμε πλήρως από τα δεδομένα αυτά. Μεταξύ άλλων δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα, υπήρχε κατακαιρματισμός, δεδομένα που ερχόντουσαν από έρευνα που χρηματοδοτόταν με δημόσιο χρήμα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα. Οπότε στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι ακριβώς να διευκολύνει όχι μόνο τη χρήση αλλά και την επαναχρήση και το να μπορούμε να μοιραζόμαστε μεταξύ μας και να ανταλλάσσουμε δεδομένα, κάτι το οποίο ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της οικονομίας, η οποία εξαρτάται κατά πολύ από τα δεδομένα. Η εκτίμηση είναι ότι η Ευρώπη με αυτό το ευρωπαϊκό ανοιχτό επιστημονικό ηλεκτρονικό νέφος θα βοηθήσει πάρα πολλούς επιστήμονες και ερευνητές να μπορούν να ξαναχρησιμοποιήσουν δεδομένα. Τώρα πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την γνωμοδότηση. Επικεντρωθήκαμε σε κάποια στοιχεία που αποτελούν ε, βέβαια μέρος της αρμοδιότητας της δικιάς μας Επιτροπής. Θεωρώ ζωτική σημασίας η πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό νέφος να βοηθήσει όχι μόνο την έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και συγχρόνως να μην αφήσει απ' έξω καμία χώρα μέλος. Ιδίως όταν μιλάμε ότι δεν υπάρχει επαρκή συμμετοχή είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι κυρίως οι μικρομεσαίες, κυβερνήσεις, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να εμπλέκονται περισσότερο στην πρωτοβουλία αυτή και να αποφεληθούν από αυτή. Επίσης, η πρωτοβουλία έχει πολλές δυνατότητες για να ε, βοηθήσει σε ανάπτυξη την ψηφιακή μας οικονομία και άρα να θέσει την ήπειρό μας ε, συνολικά στον κόσμο σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό υπέρ της ε, δικιάς μας ενιαίας αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, αγαθών, υπηρεσιών και ατόμων. Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων θα μπορούσε να θεωρηθεί η πέμπτη ελευθερία της Ένωσης. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ακόμα πιο εύκολα στην εσωτερική μας αγορά. Θα έπρεπε επίσης η Επιτροπή να επωφεληθεί από τα δεδομένα που ήδη υπάρχουν και να φροντίσει τα δεδομένα αυτά να κυκλοφορήσουν μεταξύ μας χωρίς σύνορα. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πρώτα απ' όλα να επωφεληθούμε από αυτά που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας πριν επενδύσουμε σε ακριβά νέα προγράμματα. Είμαι σκιώδης η από το ΕΛΚ και για την γνωμοδότηση του FSI που θα ψηφίσουμε αύριο και διαπίστωσα ότι δεν συμμετέχουν αρκετά τα ταμεία στην ψηφιακή τεχνολογία. Ζητάω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσει τη συμμετοχή <clears throat> του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε έργα σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά. Πρέπει να έχουμε μια αγορά που όντως εξαρτάται κατά πολύ από τα ψηφιακά δεδομένα και άρα πρέπει αυτά να κυκλοφορούν. Επειδή τώρα είναι περιορισμένος ο χώρος που έχουμε στη διάθεσή μας για γνωμοδοτήσεις, θα υποβάλω και κάποιες τροπολογίες μέσα στις οποίες θα συμπεριλάβω το θέμα της κατάρτισης ώστε να αποφελθούμε ακόμα περισσότερο από το Ευρωπαϊκό Ανοιχτό Επιστημονικό Ελεκτρονικό Νέφος και θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά κάποιου ορισμούς. Τι σημαίνει να του ανήκουν κάποιου τα δεδομένα, για παράδειγμα, και διάφορα άλλα. Όπως είπε και η Βίκη, η ΙΜΚΟ γονομοδοτεί η επί τη ουσία ε, αρμόδια επιτροπή είναι ήτρε. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Με εκ μέρου των σοσιαλιστών, η Κάθριν. Κάθριν Στήλερ. Δεν μπορεί να είναι εδώ η συγκεντριά μας, οπότε έχω ένα σημείωμα. Επειδή βρισκόμαστε στην ε, ψηφιακή επανάσταση, τα δεδομένα πρέπει να κυκλοφορούν και η Σκιώδης αναφέρθηκε στην πέμπτη ελευθερία. Όντως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια έχει και την πρωτοβουλία αυτή να βοηθήσει τους επιστήμονες, τους ερευνητές και τη δημόσια δίκηση με τα δεδομένα τα οποία θα κυκλοφορούν απρόσκοπτα για να βοηθήσουμε να πετύχει ακόμα περισσότερο η ψηφιακή μας οικονομία. Υπάρχουν τρεις πυλώνες για τον τρόπο που κυκλοφορούν, αποθηκεύονται, μεταφέρονται και φυσικά και οι υπολογιστές πρέπει να τα ανταποκρίνονται. Επίσης είπαμε Όποιοι είναι είναι δικαιούχοι. Είναι επιστήμονες, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Και κατά το δικό μας ε, εισηγητή πρέπει να αποφελθούν φυσικά και οι επιστήμονες αλλά και οι πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα τα δεδομένα και σε αυτούς και φυσικά και οι επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρξει μείωση του κόστους. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες που μας ε, δίνουν όλα αυτά. Σίγουρα υπάρχουν μέχρι τώρα κάποιες βελτιώσεις με κάποιες πανευρωπαϊκές ε, δομές, με κάποιες διευκολύνσεις αποθήκευσης δεδομένων που είναι ανοιχτή στους επιστήμονες, αλλά χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες και περισσότερη χρηματοδότηση ώστε η προσβασιμότητα στα ψηφιακά δεδομένα να είναι μεγαλύτερη. Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει να βοηθήσει και τους επιστήμονες και ερευνητές και τη δημοσιοδίκηση, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και σε περιφερειακό επίπεδο μάλιστα. Διάφορα σημεία ήθελε να αναφέρει σκιώδης εισηγητήμος που είναι οι υποδομές η βεβαιότητα που πρέπει να κυριαρχεί και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στο ηλεκτρονικό νέφος και τους καταναλωτές. Τα ωφέλη για τους καταναλωτές που πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν περισσότερο το ηλεκτρονικό νέφος εκτός από τους ερευνητές και τους επιστήμονες και επίσης να αποφεληθούν τα μέγιστα και οι επιχειρήσεις. Τέλος υπάρχει και το θέμα του κατακαιρματισμού που πρέπει να προσέξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά λοιπόν είναι τα σημεία του σκιώδη συγητή μας, που βέβαια θυμίζουν πάρα πολύ αυτά που είπε και η συγγήτρια μόλις πριν. Θα συνεργαστούμε φυσικά και προσβλέπουμε και εμείς σε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Εγώ είμαι η συντονίστρια για το ECR και σας ευχαριστώ για την καλή δουλειά σας, Εύα, για αυτή τη γνωμοδότηση, για να μεγενθηθεί η ψηφιακή οικονομία. Πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές και να διασφαλίσουμε ότι υποστηρίζουμε και το υπολογιστικό νέφος. Θα πρέπει να θέσουμε τις ευρείες αρχές ε, της Ευρωπαϊκής ε, Πρωτοβουλίας για το υπολογιστικό νέφος. Ε, πρέπει να υποστηρίζουμε την καινοτομία και φυσικά τις, ε, να είναι, είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι και να έχουμε ένα περιβάλλον που να βοηθά όσους κοινοτομούν και προκειμένου ο κλάδος ε, και τα ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν ε, να κάνουν τα πράγματα σωστά. Μου άρεσαν τα όσα είπατε σε ό,τι αφορά την ελευθερία των δεδομένων και πιστεύω ότι είναι επιτακτικό να αποφύγουμε τα εμπόδια που θα δημιουργήσουν γύρω από την Ευρώπη ένα ψηφιακό φρούριο. Ο κόσμος μας είναι ένας κόσμος χωρίς σύνορα, θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας διεθνώς για να διασφαλίσουμε ότι δεν αποκόβουμε την Ευρώπη σε ό,τι αφορά στο υπολογιστικό νέφος. η πρωτοβουλία θέλει να διασφαλίσει ότι όλα τα επιστημονικά δεδομένα μέχρι το 2020 είναι εξορισμού ανοιχτά. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά εγώ, πολύ μεγάλη δουλειά όταν διαπραγματευόμουν τον ορίζοντα 2020 και πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανταλλαγής δεδομένων και της ε, προστασίας των δεδομένων και Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κανόνες της προστασίας των δεδομένων να γίνουν σεβαστοί. Όμως υπάρχει και πολύ μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει. Τώρα δούμε με, ποιες, ε, με ποιους τρόπους λεπτομερώς θα εφαρμοστούν οι κανόνες αυτοί. Έτσι λοιπόν η εφαρμογή θα συνεχίζει να πρέπει να γίνεται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι νόμιμε ανησυχίε για την προστασία των δεδομένων. Σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, στο κράτο μέλο μου πάνω από το 60% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ε, σε πρόσφατη μελέτη είπαν ότι φοβούνται ότι θα μπορούσαν να χαθούν ε, ε, ή να πληγούν πολλά δεδομένα στο υπολογιστικό νέφος και πιστεύω ότι πολλοί ανησυχούν. Ε, πρέπει να οικοδομήσουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και προτείνω εδώ κάποια διατύπωση για το πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και λέω ότι αυτό το θέμα της κυβερνοασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί καλύτερα εντό της οδηγίας, στα πλαίσια της οδηγίας για την ασφάλεια στην στον τομέα των πληροφοριών. Σας ευχαριστούμε για τη διατύπωση σε ό,τι αφορά τα πρότυπα. Όπως ξέρετε, ήταν ένα από τα θέματα που με απασχολούσαν ιδιαίτερα και συνεχίζω να εστιάζω εκεί. Πρέπει ουσιαστικά από κάτω προς τα πάνω να τίθενται τα πρότυπα σε συνεργασία με τη βιομηχανία, με τον κλάδο και με τους παγκόσμιους εταίρους. Έχω κάποιες λοιπόν τροπολογίες να προσθέσω σε μια γνωμοδότηση που είναι ήδη πάρα πολύ καλή. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην Κάια Κάλλας. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν, ο Μάρτιν Λόκαρτ είναι ο δικός μας κοιόδης, αλλά απουσιάζει. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσει την εισηγήτρια για την πλήρη εκθεσή της. Είναι γενικά καλή η έκθεση της Επιτροπής και μπορεί να προωθήσει ακόμη περισσότερο την έννοια ψηφική αγορά. Ο Μόρτεν βέβαια έχει κάποιες, ε, κάποια σχόλια στις ε, τροπολογίες του για τη χρηματοδότηση. Δεν είναι ακόμα σαφές ε, πώς γίνεται η χρηματοδότηση μικροπρόθεσμα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να υποστηριχτεί ισχυρά μέσω του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολο να εκτελεστεί από την ε, πλευρά του Άλτε λείπει μια αναφορά στην ανοιχτή επιστήμη. Είναι ε, ουσιαστικά στο επίκεντρο της στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνδέεται με, την, με τον ορίζοντα 2020. Πρέπει τα αποτελέσματα των ερευνών να είναι πιο προσβάσιμα και αυτό συνεισφέρει σε μια αποτελεσματική επιστήμη και στην κοινοτομία, στην ιδιωτική και στη δημοσία τομέα. Όλες οι πολιτικές ομάδες είναι ενωμένε σε αυτό το σημαντικό στοιχείο που ωφελεί όλους ε, τους ανθρώπους πέρα από τα σύνορα, πέρα από τις ερευνητικές κοινότητες. Πρέπει να αναφερθούμε και στην ε, φυσική υποδομή που χρειάζεται στην Ευρώπη, ε, δηλαδή γιατί πρέπει να έχουμε υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και γρήγορη συνδεσιμότητα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τους ερευνητές να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο διοικητικό άχθος και Επίσης, ε, λέμε στον ε, εισηγητή της Ήτρε ότι δεν είναι και τόσο κακή η πρόταση της Κομισιόν. Ποιος θέλει το λόγο, κάποιος από τους Πρασίνους, παρακαλώ έχετε το λόγο, Τζούλια. Πιστεύω ότι Πολλά σημαντικά τα είπε η κυρία Κάλλα. Νομίζω ακολουθεί καλή κατεύθυνση εδώ η Κομισιόν, κυρίω με το Ευρωπαϊκό Νέφο Ανοιχτή Επιστήμης. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η πολιτική να είναι συνεκτική με άλλε πρωτοβουλίε τη Κομισιόν. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ο στόχος μας να είναι να έχουμε μια υποδομή έρευνας και να επιτρέπει σε όλους όσους εμπλέκονται στην έρευνα και στους πολίτες και στους ερευνητές να ανταλλάσσουν δεδομένα, να υπάρχει απαραίτητη διαλειτουργικότητα και να λαμβάνει χωρί ανταλλαγή δεδομένων ε, με έναν τρόπο που να επιτρέπει την απαραγωγικότητα των αποτελεσμάτων. Και υπάρχει μια δέσμευση στην ανοιχτή επιστήμη και στην ανοιχτή κοινοτομία μέσω όλων των προτάσεων πολιτικής που καταθέτει η Κομισιόν, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε στην εξή κατάσταση, να παρεμποδίζεται μια καλή πρωτοβουλία είτε από πολιτικές που εμποδίζουν ή δημιουργούν δυσκολίες για την ανοιχτή πρόσβαση ή από την έλλειψη υποδομής ε, σε ό,τι αφορά τη συνθεσιμότητα. Εύελιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστούμε και για αυτό το πολύ ενδιαφέρον σχέδιο γνωμοδότησης που μα παρουσιάστηκε. Υπάρχουν εδώ κάποιες πάρα πολύ σημαντικές πτυχές, κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία, παραδείγματο χάρη στο σημείο 12, όπου αναφέρεστε στους κινδύνους, ε, σε ό,τι ε, αφορά ε, την προστασία των δεδομένων. Τώρα, Έχω μια ερώτηση για το σημείο 5. Μήπως θα μπορούσατε να μας ε, δώσετε κάποιες λεπτομέρειες γι' αυτό. Για την έκθεση Παύλοβα. Δεν μιλάμε. Μάλιστα. Συγγνώμη που ήρθα και κάπως καθυστερημένα. Θέλω να φερθώ στον παράγραφο 5. Εδώ αναφέρεστε στον ρόλο των δεδομένων ε, στην αλυσίδα αξίας, στην αξιακή αλυσίδα. Και μιλάτε και στο πώς θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα οι ευρωπαϊκές εταιρείες. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείται με αυτό. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε. Μιλάτε για μερισμό των δεδομένων. Αν μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. I'm only looking a bit strange because in my point five... Μάλιστα, αναφερθήκα στο σημείο 5. Εδώ έχουμε μία παράγραφο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Unless Μιλάτε για το σημείο 5 στην έκθεση ΙΤΡΕ. E εκεί, στην έκθεση Ήτρε, το σημείο 5 λέει ότι... Συγγνώμη, είχα λάθος κείμενο. Κοιτάξτε, αν αναφέρει το σημείο 5 στην έκθεση Ήτρε, εκεί ζητάτε να βελτιστοποιηθούν τα δεδομένα από τις ευρωπαϊκές εταιρείες και αυτό γίνεται στην επικράτεια της Ένωσης, τότε αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Κοιτάξτε, με εξέπληξε κάπως αυτό. Γιατί ουσιαστικά δεν ε, είχα κατανοήσει πως όλα αυτά συνδέονται, αλλά τώρα τα κατανόησα. Μάλιστα να ξαναδώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια, εκτός αν Κομισιόν θέλει το λόγο. Πρώτα Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη γνωμοδότησή σας και ευχαριστώ και για τα πολύτιμα σχόλια. Πολλά από αυτά που είπατε ε, τα λάβαμε υπόψη μας όταν ετοιμάσαμε την ανακοίνωση αυτή. Υπενθυμίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η πρωτοβουλία για το ηλεκτρονικό νέφος είναι να μην υπάρχει επικάλυψη, να λάβουμε υπόψη μας τι ήδη υπάρχει δηλαδή και να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τις ήδη υπάρχουσες υποδομές ή δεδομένα. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ότι ήδη υπάρχει αντί να τα φτιάξουμε όλα από την αρχή. Όσον αφορά το σχόλιο για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων, από την αρχή λάβαμε υπόψη μας ε, τους ενδιαφερόμενους με διαβουλεύσεις, με διάφορες ομάδες εργασίας, είτε πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βιομηχανία λάβαμε υπόψη τους όσο περισσότερο μπορούσαμε τα σχόλιά τους και θα συνεχίσουμε όσο προχωράει η πρωτοβουλία αυτή. Το θέμα της εμπιστοσύνης και της ιδιωτικότητας είναι πολύ σημαντικά. Και αυτό ακριβώς εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε και το σλόγγαν που χρησιμοποιούμε. Ότι πρέπει να είναι όσο ανοιχτό το νέφος όσο γίνεται και όσο κλειστό όσο πρέπει. Όσοι έχουν κάποια εμπειρία αντιλαμβάνονται ότι στα ανοιχτά δεδομένα υπάρχουν κάποιες διατάξεις και θα υπάρχουν και στο νέφος, στο ηλεκτρονικό, που λέει ότι όταν κάποια προγράμματα δεν πρέπει να είναι ανοιχτά για λόγους ιδιωτικότητας ή οτιδήποτε άλλο, θα γίνεται. Άρα δεν είναι ένα πλήρως ανοιχτό. Αυτά Λαμβάνονται υπόψη λοιπόν. Και αυτά τα στοιχεία νομίζω θα σας βοηθήσουν να συντάξετε και την τελική σας γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ και για την επικοδομητική σας στήριξη. Η συγήτρια. η Εύα Πανόβ. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχαν στη σημερινή συζήτηση. Χαίρομαι που ταυτίζεται η προσέγγισή μας. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι η γνωμοδότησή μου θα επικεντρωθεί όσο γίνεται περισσότερο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της ΙΜΚΟ. Προσβλέπω στις τροπολογίες σας και αυτό που είπα στην αρχή είναι ότι επειδή περιοριζόμαστε στις γνωμοδοτήσεις μας, δεν μπόρεσα να συμπεριλάβω κάποια σχόλια όπως αυτά που ακούστηκαν για το ανοιχτό επιστημονικό ηλεκτρονικό νέφος και κάποια άλλα. Οπότε περιμένουμε τις τροπολογίες και προσβλέπω σε συνεργασία με τους σκιώδες εισηγητές. 13 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Μην το ξεχνάτε αυτό. Θα βοηθούσε πολύ. Και επίσης, ελπίζω, η Ήτρε να συμπεριλάβει όσο γίνεται περισσότερες από τις παρατηρήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ενωμένη κατά του προστατευτισμού. Το επόμενο σημείο στην ημερησία διάταξη έχει να κάνει με την έκθεση Μακλάρκιν. Μάλιστα. Τέλεια. Πολύ ωραία να έχουμε για κάποιον από τους κυρίους στην Επιτροπή εδώ σήμερα. Γιατί νόμιζα ότι θα ήταν η μέρα των γυναικών σήμερα. Σημείο 7. Ε, Συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων εν ώψη των μεταβαλλόμενων συνθήκων της αγοράς. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα μιλήσουμε για τα πολεμικά βίντεο. Και τώρα, η κυρία Μακλάρκιν, βάσει του κανόνα 53, εκδίδει μια γνωμοδότηση για την Επιτροπή Κολτ, ε, όπου έχουμε συνεισηγήτριες, την Πέτρα Κανούβα και τη Σαμπίν. Βερχέιεν, παρακαλώ, θα σας δώσω το λόγο για να παρουσιάσετε την έκθεση. Δυστυχώς η ΑΜΑ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Εγώ θα παρουσιάσω την έκθεση. Έτσι λοιπόν η οδηγία για το οικογνωστικά μέσα αποτελεί ε, ουσιαστικά ε, ένα πλαίσιο ισχυρό που μπορεί να καλύψει τις πολιτιστικές ευαισθησίες των κρατών μελών ενώ ουσιαστικά ε, παρέχει το, το ελάχιστο δυνατό άχθος. Έχουμε ουσιαστικά τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο που ουσιαστικά καθιστά αναγκαία να τροποποιηθεί η οδηγία για τα ακουστικά μέσα και αυτή η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή ε, θα πρέπει να απασχολεί αυτή την Επιτροπή, εντάξουμε τις υπηρεσίες ε, αυτές ε, στην οδηγία υπηρεσιών οπτικοστικών μέσων για να αντιμετωπίσουμε την υποκίνηση μίσου, Εδώ θέλουμε στη, να συμπεριλάβουμε τις γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίε εδώ θέλουμε ουσιαστικά να θέσουμε τέλος στη διάκριση στους μη ευρωπαϊκούς χρήστες τώρα, κατά την άποψή μου υπάρχουν καλύτεροι τρόποι όπως ο έλεγχος των γονεών και το αλφαβητισμός στα μέσα για να προστατεύσουμε τους καταναλωτέ. Επίσης ε, θα έχουμε και το θέμα εδώ της ευθύνης των πλατφόρμων που σήμερα είναι περιορισμένοι που αυτά τα σχέδια οργανώσει θα μπορούσαν να καθιστούν υπεύθυνε για το περιεχόμενο παρόλο που δεν έχουν συντακτική ευθύνη ούτε καν ξέρουν ότι έχει ανέβει ε, στην ιστοσελίδα τους. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν είχε προτείνει τους κανονισμούς ε, στη, ότι θα πρέπει να υπάρχει μέγιστη προσέγγιση εναρμόνισης αν υπάρξει η χορήγηση δυνατότητα των κρατών μελών να ε, νομοδοτήσουν για ε, τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικό καθεστώς στα κράτη-μέλη και αυτό θα ήταν πολύ δύσκολο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την νέα αγορά. Το θέμα της διατήρησης της αρχής της χώρας προέλευσης είναι η ραχοκοκαλιά αυτού του κανονισμού και εμείς ε, σε οποιαδήποτε, προσε... οποιαδήποτε μετακίνηση προς ε, την προσέγγιση της χώρας προορισμού θα αποδυνάμωνε περαιτέρω την αρχή της χώρας προέλευση και θα σε ολιστηρό έδαφος. Έτσι λοιπόν γι' αυτό το λέγω για να μην αναφέρω και ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ε, για να δείξουμε ότι δεν ε, θα αυξάνονταν οι επενδύσει, ε, Αποσύρονται οι εισφορέ τα τέλη είναι σημαντική η προστασία των καταναλωτών και για την οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό η δική μας επιτροπή να δεσμευτεί στο να διατηρήσουμε την αρχή της χώρας προέλευσης. Η οδηγία EVMS πρέπει να συνεχίσει να υπερασπίσει τις ε, ελεύθερες αξίες της αγοράς. Ε, έχουμε ε, κάποιες, ε, παραδείγματος χάρη, απαιτήσει όπως είναι η προβολή ε, και η αποκάλυψη του περιεχομένου που δεν συνάδουν με τις αρχές αυτές, οποιαδήποτε κίνηση προς τον προστατευτισμό ε, ουσιαστικά δεν θα εξυπηρετούσε αυτό που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση την ευρεία αγορά. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι για το περιεχόμενο που παράγουμε και θέλουμε ουσιαστικά τον ανταγωνισμό και εδώ βλέπουμε τη μεγιστοποίηση των επενδύσεων και την δυνατότητα να παράγουμε περισσότερο ποιοτικό περιεχόμενο. Έτσι λοιπόν, ενώ ευνοούμε μια προσέγγιση ε, της αγοράς ε, στις περισσότερες ε, περιπτώσεις ο εισηγητής θέλει 12 λεπτά ανά ώρα για τις εμφυμίσεις το, 20, το όριο της 24, των 24 ωρών μπορεί να βλάψει τους καταναλωτές. Επίσης το όριο, αν αυξήσουμε το όριο στις 24 ώρες, θα έχουμε μείωση των εσόδων από τις διαφημίσεις και όχι αύξηση. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην διευρύνουμε ουσιαστικά το πεδίο πέρα από την επιθυμητό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η αρχή της χώρας προέλευσης παραμένει κέριο στοιχείο αυτής της οδηγίας.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 περιλαμβάνονται στο σχέδιο γνωμοδότησης της εισηγήτης με το οποίο συμφωνούμε και συμφωνούμε ότι το πεδίο εφαρμογής δεν πρέπει να περιορίζεται και η αρχή της χώρας προέλευσης πρέπει να διαφυλαχθεί. Επίσης, συμφωνούμε με μια προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά τις πλατφόρμες video sharing από τη μια λοιπόν πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνουμε δυνατότητες στους καταναλωτές να αναφέρουν ε, περιεχόμενο, αλλά πρέπει αυτό να γίνεται λογικά και δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη το θέμα της ηλικίας. γιατί είναι σημαντικό να βλέπουμε ποια είναι τα κοινά και ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο γραμμικό και μη γραμμικό περιεχόμενο. Στη Γερμανία είχαμε παραδείγματα με χρονοθυρίδες που βάζαμε στο διαδίκτυο. Που βέβαια δεν έχει πάντα νόημα γιατί κάπου στον κόσμο θα είναι πάντα μετά τις 10 το βράδυ. Επίσης έχουμε επιφυλάξεις για την απορρίθμιση της διαφήμισης στις γραμμικές αναμεταδόσεις. Και για το θέμα των πλατφορμών video sharing είναι πολύ σημαντικό οι ορισμοί να είναι σωστοί. Άλλο είναι η υπηρεσία που έχει κάποια ευθύνη περιεχομένου και άλλο είναι οι πλατφόρμες video sharing που δεν έχουν τέτοια ευθύνη. Οπότε η ποσόστοση εκεί δεν εφαρμόζεται. Νομίζω ότι το σχέδιο βέβαια έκθεσης από την Επιτροπή Πολιτισμού μπορεί κανείς να το δει έτσι, αλλά είναι σημαντικό να διευκρινιστεί γιατί η ποσόστοση σε τέτοιες πλατφόρμες δεν έχει νόημα. Εκεί που δεν συμφωνούμε είναι στο ρόλο των ρυθμιστών. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο παράγοντας ανεξαρτησίας και για τις αναμεταδόσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να υπάρχει ποικιλομορφία και δημοκρατία στα μέσα αναμετάδοσης. Και εδώ λοιπόν θα υποβάλουμε τροπολογίες. Πάντως πιστεύουμε ότι γενικά είναι πολύ σημαντικό για την ΙΜΚΟ να ολοκληρώσει γρήγορα την γνωμοδότησή της. Και είναι εφικτό. Γιατί έτσι στις διαπραγματεύσεις οι ανησυχίες της Επιτροπής μας για την εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα ληφθούν περισσότερο υπόψη. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ υπάρχει κάποιος. Όχι. Ωραία. Παρακαλώ, κυρία Χετ, τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Δεν ακούγεται κυρία Χεντ. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο της κυρίας Head. Δεν την ακούμε την κυρία Head. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο της. Μπορείτε να αρχίσετε και πάλι. Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Το μικρόφωνο της κυρίας Head δεν λειτουργεί. Το μικρόφωνο είναι το πρόβλημα. Το μικρόφωνο. Μπορείτε να αλλάξετε θέση γιατί δεν λειτουργεί το μικρόφωνο σας. Γιατί εμεί μεν σας ακούγαμε, αλλά οι διερμηνείς δεν σας άκουγαν. Ωραία, τώρα με ακούτε. Καλώς. Τώρα λειτουργεί. Ναι, ευχαριστώ. Αρχίζω και πάλι. Θα αρχίσω και πάλι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή πρέπει να σας πω ότι ήμουνα παρούσα την προηγούμενη φορά όταν συζητήσαμε και υπάρχουν κάποια στοιχεία εδώ τα οποία μπήκαν στην πάντα. Όπως και την προηγούμενη φορά, νομίζω. Κάποιες από τις υπηρεσίες αυτές είναι πολύ σημαντικές σε καθημερινή βάση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε τα πράγματα με τα μάτια του καταναλωτή. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο για τον καταναλωτή ότι προστατεύεται από τις ρυθμίσεις αυτές. Κυρίως τα παιδιά. Για τους θετές αυτούς τους ανήλικους οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται από τη διαφήμιση, προγράμματα κλπ. Πρέπει λοιπόν να προστατεύουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Και όσον αφορά την ε, πολιτική εκστρατεία πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας. Υπάρχει περιοριστική πολιτική στη Σουηδία για τα ενοπνευματόδη, το οποίο είναι πάντα παρόντα. Είναι συμφέρον όλων μας να προστατεύσουμε τα παιδιά και την κοινωνία από διαφημίσεις για ενοπνευματόδη ποτά, για παράδειγμα. Να δούμε λοιπόν τι ισχύει όσον αφορά τη διαφήμιση των ενοπνευματοδών και το ίδιο και για τα προϊόντα καπνού. Οι καταναλωτές πρέπει να προστατεύονται με έναν σε ένα ευρύ πλαίσιο. Εμείς λοιπόν εδώ πρέπει επίσης να φροντίσουμε να αποφύγουμε την όθηση στο έγκλημα, στη βία, τη ρητορική, μίσους. Η κοινωνία το έχει καταλάβει και μας το λέει και μας το ξαναλέει ότι αυτά που θέλουμε για τα οπτικουστικά δεν πρέπει βέβαια να περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να βρεθεί η σωστή ισορροπία. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Θα καταθέσουμε και εμείς τροπολογίες λοιπόν. Και η συγκήτρια σίγουρα θα συγκεντρώσει τους κοιόδης συζητητές να συναντηθούμε και να ακούσουμε ένα τον άλλον τι έχουμε να πούμε. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Εκ μέρους του Μόρτον θα μιλήσω εγώ. Θέλει να αναφέρει κάποια σημεία καλωσορίζει την ισορροπημένη έκθεση Μακλάκιν για τις ποσοστώσεις. Λέει ότι πρέπει να το κοιτάξουμε και να βρούμε μια εναλλακτική, γιατί λέει ότι δεν λύνουν το πρόβλημα. Είναι σαφές πώς θα βοηθήσουν οι ποσοστώσεις. Και γενικά είναι υπέρ συνεργασία μεταξύ των ε, μεταδοτών προγραμμάτων και των αρχών. Έπειτα και για την οικονομική χρηματοδότηση δεν βλέπει να υπάρχει εδώ λύση. Επειδή έρχεται από μικρή χώρα μέλος, βρίσκει ότι είναι σημαντικό η πρόταση αυτή να καλύπτει όχι μόνο τις μεγάλες χώρες μέλη, αλλά και τις μικρότερες, να φροντίζει να τις προστατεύει και κυρίως τις λιγότερο μιλούμενες γλώσσες. Τέλος, εδώ τίθεται θέμα συνόρων η, η, τα ανοιχτά σύνορα, η ελευθερία έκφραση στο διαδίκτυο, ε, να υπάρχει ελεύθερη ε, κυκλοφορία, ναι, αλλά να μην υπάρχει διαρροή εγκεφάλων. Τώρα θέλω και εγώ να πω κάτι, δεν ξέρω τώρα ή μετά. Τώρα, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω την Πρόεδρο ίσως. Έχουμε κάνει τίποτα για τη σύγκρουση συμφερόντων με τον εισηγητή στην Επιτροπή Πολιτισμού, γιατί προφανώς και στηρίζει τα συμφέροντα του κλάδου. Οπότε δεν ξέρω πώς πρέπει να ρωτήσουμε τη διάσκεψη των Προέδρων από αυτού, να αποφασίσει. Επί της ουσίας τώρα. Οι πλατφόρμες video sharing Εδώ το πράγμα έχει ως εξής. Καταλαβαίνω αυτό που λέει και ότι πρέπει να καταλάβουμε πρώτα απ' όλα συμπεριφορές, εισηγήτρια μάλλον, σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά η αυτορύθμιση έχει φανεί, η, η συνρύθμιση, ότι λειτουργεί καλά. Και μειώνεται η παιδική πορνογραφία, δεδομένου ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται τόσο γρήγορα. Και όταν εμείς ετοιμάσουμε τη δικιά μας τη ρύθμιση, μπορεί αυτά που προβλέπουμε να είναι ξεπερασμένα, γιατί η τεχνολογία μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα από εμά. Πάντως δεν πιστεύω ότι η πρόταση της Επιτροπής ή το θέμα της όθησης στη βία ή η ρητορική μίσους. Ναι, πρέπει να υπάρχει μια πολιτική, αλλά δεν θα την αποφασίζουν οι επιχειρήσεις. δεν πρέπει να υπάρχει περιορισμός ελευθερίας ε, έκφρασης, άρα πάλι σωστή ισορροπία. Τώρα, η, η συγκήτρια προτιμάει κώδικες δεντολογίες σε εθνικό επίπεδο. Αν όμως θέλουμε εμείς, οι εταιρείε να είναι παρούσες πανευρωπαϊκά, τότε πρέπει να ενθαρρύνουμε και την ανάπτυξη κωδικών δεντολογίας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο. Τένις. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα. Δεν άκουσα τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εγώ. Γιατί εξακολουθούμε να εξετάζουμε λεπτομερώς τα εγγραφά στην ομάδα μου. Είχαμε τονίσει κάποια θέματα, κυρίως το θέμα της διαφήμισης, ε, των διαφημίσεων που απευθύνονται στα παιδιά. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι όταν μιλάμε για τις ε, υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, αν αφήσει τα πάντα στην αγορά, αυτό σημαίνει πιθανότατα ότι δεν ε, προσφέρει αρκετές υπηρεσίες και πρέπει να δούμε και το θέμα των μειονοτήτων, ε, παραδείγματο χάρη, υπηρεσίες που αφορούν τη γλώσσα και αυτό που η Κομισιόν σε σχέση με τα ευρωπαϊκά έργα. Όμως, ε, νομίζω ότι η συγγήτρια έχει πάρα πολύ εμπιστοσύνη στην αγορά. Σίγουρα θέλουμε να έχουμε κάποιες εγγύσεις ότι ό,τι δεν μπορεί να ρυθμιστεί από την αγορά θα μπορεί ουσιαστικά να καλυφθεί από όσους θέλουν να αναλάβουν και να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Στο παρελθόν ήμουν και σκιώδης για την οδηγία των οπτικοκουστικών μέσων και κάποια θέματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση, νομίζω ότι ισχύουν και για την έκθεση αυτή. Υπάρχουν άλλοι που θέλουν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για να είμαι ειλικρινής, η πραγματική συνεισφορά τη αναθεωρημένη οδηγία για τι υπηρεσίε οπτικών μέσων είναι περιορισμένη. Προφανώ έχει νόημα στο πλαίσιο τη ε, του θεματολογίου της ενίας ψηφιακής αγοράς, αλλά εγώ θα περιμένα κάτι πιο φιλόδοξο και λιγότερο περιοριστικό. Το ότι θα εισαχθούν έλεγχοι ηλικιακοί είναι κάτι καλό, συμφωνώ με τους προλαλήσατες και επίσης ε, προγράμματα ε, τα οποία ε, ουσιαστικά απευθύνεται στους ανηλίκους θα πρέπει να περιστούν σε περίπτωση που μιλάμε για ανηλίκους με Όμως εδώ θα πρέπει να δούμε ότι το ίντερνετ διαφέρει από την τηλεόραση. Το να προσπαθήσουμε να εφαρμο... αντί να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες που ισχύουν στην τηλεόραση για το ίντερνετ, ίσως θα πρέπει ουσιαστικά να περιορίσουμε ε, τους κανόνες. Ε, το να βρούμε την σωστή ισορροπία είναι πάντα κάτι δύσκολο ουσιαστικά ποιο είναι το σωστό ποσοστό ευρωπαϊκού περιεχομένου στην τηλεόραση, 20%, 30%, 10% κανένα στόχος. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ε, στόχος ε, για κάποιους, αλλά νομίζω ότι κάποιοι διαφωνούν. Θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί σε ό,τι αφορά ε, και το θέμα των εθνικού περιεχομένου. Η η υποχρεωτική προσβασιμότητα πρέπει να συμπεριληφθεί στην πρόταση. Μας είπε η Κομισιόν ότι θα ισχύσει κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε τελικά ότι δεν ισχύει. Um, ευχαριστώ. Συγγνώμη. Ευχαριστώ, Βίκη. Συγγνώμη που καθυστέρησα κι εγώ. Για ένα λεπτό θα ήθελα να πω και εγώ κάτι για την προσβασιμότητα, όσα είπε η συνάδελφος δηλαδή. Συζητήσαμε αυτό το θέμα με πολλούς συναδέλφους πριν από αυτή τη συνεδρίαση. Λείπει πάρα πολύ σε αυτή την νομοθετική πρόταση. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι όχι μόνο η δυνατότητα μεταφοράς που τη συζητήσαμε στην Επιτροπή μας, η φορητότητα, αλλά και η προσβασιμότητα Πρέπει επιτέλους οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα, σε ψηφιακό περιεχόμενο σε άλλες χώρες. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Αυτό λείπει στην έκθεση αυτή και μέσω των τροπολογιών μας ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. I want ask, make couple Ήθελα να κάνω κάποια σχόλια καταρχήν. Και άκουσα πολύ προσεκτικά αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ στο όσο είπε η κυρία Κάλλας. Δηλαδή, να διασφαλίσουμε ότι δεν είμαστε υπερβολικά περιοριστικοί σε ό,τι αφορά τα θέματα της ελευθερίας του λόγου, της ελευθερίας έκφρασης. Φυσικά θα πρέπει να δούμε τα θέματα προστασία των παιδιών, τα θέματα ρητορική του μίσου, αλλά αρχίζουμε τώρα να είμαστε πολύ περιοριστικοί για το τι επιτρέπεται να παρακολουθούν οι άνθρωποι, τότε χάνουμε πάρα πολλά από τις ελευθερίες των μέσων. Έτσι λοιπόν, Κάια, θα ήθελα να μου πεις ε, τι είδους και σκέφτεσαι να καταθέσεις και να σε υποστηρίξω σε αυτό. Είναι πολύ δύσκολος ε, τομέας, αλλά άκουσα κάποιοι να το περιγράφουν αυτό ουσιαστικά ως ε, το τέλος της συντακτικής ποιότητας, δηλαδή σε σχέση με το να αποφασίσουμε τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι αποδεκτό να δημοσιεύει κανεί. Και αν αρχίσουμε εμεί να είμαστε πάλι πολύ περιοριστικέ πολιτικοί για το τι είναι αποδεκτό, τότε ουσιαστικά λέμε και τι. Ουσιαστικά, σε αντίθεση μάλλον με το τι δεν είναι αποδεκτό. Έχω και ένα θέμα σε ό,τι αφορά αυτά τα τέλη, όπως έχουν κατατεθεί από την Κομισιόν. Ξέρω ότι η συγγήτρια προσπάθησε να το αλλάξει όμως αν έχουμε νέα αγορά στις υπηρεσίες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν άνθρωποι υπηρεσίες σε διάφορα κράτη-μέλη και δεν αρχίσουμε να λέμε αν ναι, εσύ θα προσφέρεις υπηρεσίες στη δική μου χώρα, εγώ θα βάλω πρόσθετο τέλος ή φόρο σε σένα που θα πάει σε ένα ταμείο που μόνο εγώ θα χρησιμοποιώ για να υποστηρίζω τη δική μου εγχώρια βιομηχανία. Αυτό νομίζω ότι είναι εντελώ παράλογο. Τώρα, αν ε, λέμε όπως κάνουν κάποια κράτη-μέλη ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε το εθνικό περιεχόμενο λέγοντας ότι θα σας δώσουμε φορολογικές ελευθερίνσεις και όλοι μπορούν παραδείγματο χάρη να συμμετέχουν αν δεν θέλουν ε, να κάνουν κάποιες ταινίες στο Βέλγιο, στη Λετωνία μπορεί παραδείγματο χάρη οποιοδήποτε να θέλει να έρθει στο Βέλγιο και να του προσφερθούν φορολογικέ ελευρήσεις ή φορολογικά κίνητρα, εντάξει, αλλά αν βάζει μια φορά σε μια αλλοδαπή εταιρεία και λε, αυτό πηγαίνει σε ένα ταμείο και θα το χρησιμοποιήσω αυτό μόνο για να επιδοτήσω το δικό μου επιλεγμένο εθνικό περιεχόμενο, δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια προσέγγιση που αρμόζει στην ίδια αγορά. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρούμε εδώ μια διαφορετική διατύπωση για το πώς μπορούμε να έχουμε ένα θεμητό ανταγωνισμό, ενώ θα υποστηρίζουμε ταυτόχρονα και την εγχώρια πολιτιστική παραγωγή. Συγγνώμη, ήθελα απλώς να τα πω. Η Κομισιόν, παρακαλώ. Θέλεις να επανέλθεις, ε, Νταν. Ως Νταν, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω σε ένα άλλο θέμα. Τώρα είναι η προσωπική άποψη. Φυσικά θα τα περάσω όλα αυτά ποτέ στον εισηγητή. Από τη δικιά μου οπτική συμφωνώ με αυτό που υπόθηκαν ότι πρέπει να μειώσουμε το περιεχόμενο το οπτικοακουστικό και όχι να το αυξήσουμε. Όσον αφορά από την πλευρά του καταναλωτή, πρέπει να υπάρχουν σωστοί κανόνε για του ανήλικου και τα παιδιά, πρέπει να του προστατεύσουμε και να αντιμετωπίσουμε και τη ρητορική μίσου. Αλλά αυτό που έχει κάνει το ίντερνετ με τις πλατφόρμες ε, καταζήτηση on demand, τώρα μπορούν απλά οι καταναλωτέ να κλείσουν το δέκτη, να δουν κάτι άλλο, να δουν οτιδήποτε θέλουν οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και δεν χρειάζεται να περιμένουν καν. Αυτό λοιπόν που προτείνεται δεν έχει λογική. Έχουμε ε, δεν χρειάζεται να δούμε το 20% από όλα αυτά. Αν υπάρχουν κάποια που, ε, κάποιες που δεν θέλουν να δουν, θα τις δουν άσχετα με τα ποσοστά, με τις ποσοστώσεις. Τώρα, όσον αφορά τα VSP, δεν έχουν έλεγχο, άρα δεν μπορούν να έχουν υποχρέωση για τοποθέτηση προϊόντων ε, όσον αφορά τις πλατφόρμες αλλαγή βίντεο, τα VSP. Επομένως θεωρώ ότι έχουμε κάποια θέματα που θα πρέπει να τα επιλύσουμε. Θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε αυτούς τους κανόνες ενδεχομένω σε, μια, ε, σε ένα ενισχυμένο καταναλωτικό περιβάλλον. Όμως ε, αυτό που έχει κάνει το ίντερνετ και πρέπει να το λάβουμε είναι ότι έχει ενισχύσει, έχει δυναμώσει τους ε, καταναλωτές. Και όλα τα υπόλοιπα φυσικά θα τα διαβιβάσω στον εισηγητή Όμω βλέπω ότι έχουμε ξεκινήσει να έχουμε μια κοινή θέση και επομένω είμαι και ευχαριστημένο με αυτά που βλέπω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για να Έχουμε μια απάντηση στην ερώτηση ΚΑΕ για τη σύγκριση συμφερόντων. Έχουμε εδώ δύο συγγητές και από ό,τι κατάλαβα αυτό το θέμα τέθηκε και πώς να το πω ευγενικά δεν υπήρχε πλειοψηφία εντός των ομάδων για να υποστηρίξουν να πάμε παραπέρα σε αυτό το θέμα. Thank you uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για το σχέδιο γνωμοδότησης. Διαβάζοντας την γνωμοδότηση και ακούγοντας και εσάς, ε, βλέπω ότι έχουμε κοινούς στόχους. Απλώς έχουμε βρει φροντικές λύσεις ξεκινώντας με τις ε, VSP πλατφόρμες. Πρέπει να βρούμε μια ε, χρησιτομένα μέσα στην προστασία και την ελευθερία του λόγου και να γνωρίσουμε το γεγονός ότι ε, δεν υπάρχουν όλες τις δυνατότητες. Η πρόθεσή σας να, να προωθήσετε την αυτορύθμιση ή την αποκοινού ρύθμιση θα ήθελα σε αυτό να σας πω απλώς ότι νομικά αυτό δεν είναι εφικτό γιατί πρόκειται περί οδηγίας. Την ώρα που την ε, σχεδιάζαμε ήδη το είχαμε σκεφτεί αυτό και όταν έχουμε λοιπόν μια οδηγία δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τα κράτη, μέλη, ποια θα είναι τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους ε, ενθαρρύνουμε ώστε να υπάρχει συνομοθέτηση αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε απλώς να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο επιλέξαμε αυτήν την οδό. Όσον αφορά τη χώρα καταγωγής, θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι η βασική μας γραμμή και γι' αυτό στον μηχανισμό απόκλησης έχουμε αυξήσει το, τη χρονική προθεσμία γιατί έχουμε ήδη αντιμετωπίσει περιστάσεις όπου χρειάστηκε να θετήσουμε αποκλήσεις τέτοιου είδου και είναι πολύ δύσκολες αυτές οι αποφάσει. γιατί πρόκειται περί μιας απόκληση μια θεμελιώδη ελευθερία, κάτι που πρέπει να αξιολογήσει η Επιτροπή και κάθε φορά που ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία έπρεπε να καταφύγουμε στην επίγουσα διαδικασία, επίγουσα διαδικασία, γιατί θα χρειαζόταν πολύ χρόνο να έπρεπε να λάβουμε υπόψη όλε τι διαβουλεύσει. Τώρα υπάρχει διαβούλευση στο πλαίσιο του έργα γιατί η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη τους είναι πολύ σημαντική για εμάς και γι' αυτό προτείνουμε την ε, επέκταση της ε, προθεσμίας. Όσον αφορά τις ποσοστάσεις ε, στους παρόχους on demand, σε αυτό το σημείο θα συμφωνήσω ότι το να έχουμε ποσόστοση δεν είναι ιδανική λύση. Συγκεκριμένα για τις υπηρεσίε on demand. Γιατί μπορεί να έχουμε μία ποσόστοση της τάξης του 20%. Αλλά έτσι μπορούμε να πάμε στο Netflix ε, και να δούμε και το υπόλοιπο 80%. Άρα η ποσόστοση δεν θα είναι αποτελεσματική και γι' αυτό στην πρότασή μας συνδυάζουμε μια μικρή ποσόστοση, το 20% είναι μια χαρά παράλληλα με την υποχρέωση προώθησης. Αυτό που τελικά είναι αποτελεσματικό είναι η πρόθεση συγκεκριμένου ευρωπαϊκού ε, περιεχομένου όσον αφορά τις ε, εισφορές θα πρέπει να λευκάνουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Την 1η Σεπτεμβρίου η Επιτροπή υιοθέτησε μια απόφαση για ένα σύστημα εισφορών σύμφωνα με την οδηγία για τις υπηρεσίες πρωτοκοστικών μέσων Επέβαλε λοιπόν εισφορές σε όλους τους παρόχους που ε, έκαναν διανομές σε συγκεκριμένες χώρες και οι ανταγωνιστές σε μια συγκεκριμένη αγορά υπόκεινται στις ίδιες ε, οικονομικές υποχρεώσεις. Όμως ε, η απόφαση αυτή να εναπόκειται στην δεκτική ευκαιρία των κρατών μελών. Δεν μπορεί να επιβληθεί. Γι' αυτό θέλουμε να είμαστε βέβαιοι όπως είπε και η πρόεδρος, δεν θέλουμε να κατευθύνουμε σε μια ε, κατεύθυνση που δεν θα μας άρεσε πραγματικά. Αυτό που θέλουμε να προωθήσουμε την ε, χώρια παραγωγή, την εσωτερική παραγωγή και να είναι παράλληλα ε, συμβατά όλα αυτά με τους κανόνες ώστε να υποφεληθούν όλοι αυτοί που έχουν συνεισφέρει στην παραγωγή του περιεχομένου είτε είναι από άλλη χώρα είτε είναι από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτιμούμε λοιπόν να έχουμε αυτή την διευκρίνηση στο νομικό κείμενο ότι γίνονται σεβαστοί οι κανόνες, οι νόμοι, ώστε να είμαστε ε, βέβαιοι και σαφείς ως προς την νομοθεσία. Τώρα, όσον αφορά τη διαφήμιση, αναφέρθηκε σήμερα ότι χρειάζεται να έχουμε απορρίθμιση Υπάρχει ένα πεδίο εφαρμογή ε, όπου μπορεί να είναι δυνατή αυτή η απορρίθμιση και θα δώσει περισσότερη ευελιξία στους, ε, στα κανάλια. Γιατί το 20% που ισχύει μέχρι σήμερα δεν είναι απαραίτητο. Γιατί όταν εμείς βλέπουμε τηλεόραση, δεν υπάρχει κατάχρηση στις διαφημίσεις, τότε πολύ απλά παίρνουμε το τάμπλετ μας, όπου δεν υπάρχουν φυσικά διαφημίσεις. Ένας ε, ένα κανάλι που θα καταχρηστεί αυτό το 20% φυσικά είναι σαν να αυτοκτονεί γιατί θα χάσει το κοινό του. Άρα θεωρούμε ότι πλέον δεν υπάρχει ανάγκη να επιβάλλουμε αυτή την υποχρέωση. Αυτή είναι η λογική μας. Τώρα στην προσβασιμότητα θα πρέπει να επαναλάβω αυτά που είπε ο Επίτροπος Oettinger πολλές φορές. Αν οι συνομοθέτες καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες προσβασιμότητας θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ, τότε φυσικά θα είμαστε πρόθυμοι να το συμπεριλάβουμε. Όμως τεχνικά σε αυτό το στάδιο η Επιτροπή δεν μπορούσε να υποστήριξει κανόνες σε δύο διαφορετικά νομοθετικά ε, εργαλεία. Ευχαριστώ πολύ. Would the like to come back in for comment, or Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Θα σας δώσουμε το λόγο για τα σχόλια. Μάλιστα. Θα τα διαβιβάσω όλα αυτά στην εισηγήτρια και φυσικά είναι υπομονή να συνεργαστεί με όλους για να έχουμε τελικά μια καλή γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ προθεσμία κατάθεση τροπολογιών στις 17 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η επόμενη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Ε, Ωραία. Τώρα θα προχωρήσουμε στην ε, στα μέσα για καλύτερη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών θα έχουμε μια παρουσίαση από την Κομισιόν. Δεν ξέρω. Dan είναι το όνομά σας για το εργαλείο μελέτης αντικτύπου για τους καταναλωτές και για τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών. Θα σας δώσω λοιπόν αμέσω το λόγο. Μόλις έχουμε και τις διαφάνειες διαθέσιμες. Oh, Μάλιστα, στην οθόνη είναι η διαφάνεια. Σας ευχαριστώ. Και παρακαλώ Όποιο φύγει σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεστε για του καταναλωτέ. Θα σημειώσουμε το όνομά σα. Okay. Good. I've taken the name. Μάλιστα. Το σημείωσα και θα τον φέρουμε και στη συνεδρίες των συντονιστών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, Νταν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ και για το προμόσιο για την πρόθεση σας. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να σας ε, παρουσιάσω δύο σημεία. Καταρχήν ε, το μήνα καπιδάσεων καταναλωτικών αγαθών για το 2016 και κατόπιν το εργαλείο μελέτης αντικτύπου για τους καταναλωτές. Να σας επενθυμίσω το περιεχόμενο πίνακας επιδόσεων θεσπίστηκε το 2008 και αποτελεί τρεχοκοκολιά των ε, αποδεικτικών στοιχείων για τους καταναλωτές που συλλέγει και αναλύει η Κομισιόν. Υπάρχουν δύο είδη πίνακα επιδόσεων, αφορούν ε, να παρακολουθούν τα αποτελέσματα στην ε, αγορά. Έχουμε τον πίνακα για ε, Τι καταναλωτικέ συνθήκες. Το τελευταίο δημοσιεύτηκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Αξιολογεί το καταναλωτικό περιβάλλον στα κράτη-μέλη. Έχουμε τρεις διαστάσεις, γνώση και εμπιστοσύνη, επιβολή και συμμόρφωση και ε, καταγγελίες και διευθέτηση διαφορών και επίσης εξετάζει την ολοκλήρωση της αγοράς λιανικής διασυνοριακά και ουσιαστικά πώς ε, προωθείται το ηλεκτρονικό εμπόριο. Και κατόπιν έχουμε τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών. Το κύριο θέμα αυτής της παρουσίαση. η τελευταία προσθήκη έγινε το Σεπτέμβριο φέτος ουσιαστικά εξετάζει την επίδοση των καταναλωτικών αγορών από μια καταναλωτική σκοπιά σε πολλές διαστάσεις, ε, τη συγκρισιμότητα, την επιλογή, την εμπιστοσύνη ε, και ουσιαστικά τις το τι αναμένει ο καταναλωτής. Είχαμε πλήρη μεθοδολογική αναθεώρηση και διαβουλευτήκαμε με διαφερόμενα μένη και με διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν. Είχαμε και επιστημονική υποστήριξη από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο και ήμασταν και σε επαφή με τη γραμματεία ΙΜΚΟ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Και αυτό κατέληξε σε μια σειρά μεθοδολογικών βελτιώσεων. Τώρα, θα αναφερθώ στο τελευταίο πίνακα επιδόσεων καταναλωτικών αγαθών. Για να ξεκινήσω, να σας πω ότι δίνει μια επισκόπηση για το πώς βιώνουν ε, οι πολίτες τη λειτουργία των καταναλωτικών αγορών σε Κύριε αγαθά και υπηρεσίες σε βάση δεδομένου που συλλέχθηκαν το 2015 βασίζεται στο πέπτο κύμα μιας μεγάλης έρευνας που ρώτησε τους καταναλωτές με συγκεκριμένες πρόσθετες εμπειρίες για το ποιες ήταν οι αντιλήψεις τους ό,τι αφορά όλες αυτές τις αγορές, καλύφθηκαν όλα τα κρατημέλη, Ισλανδία και Νορβηγία και βλέπετε κάποιες πληροφορίες για το δείγμα. Είχαμε 500 ανά αναγορά και αναχώρα, γενικά με την εξαίρεση τεσσάρων χωρών. Βλέπουμε ότι αφού συλλέχθησαν το 2015 δεδομένα, χρησιμεύουν για να παρακολουθούμε την επίδοση των αγορών και να έχουμε μία επισκόπηση της αξιολόγησης της λειτουργίας ε, των αγορών πριν να ε, συγγνώμη, πριν να τεθούν σε εφαρμογή κάποια μέτρα της Επιτροπής Juncker. Καλύπτονται 42 αγορές στην έκδοση του 2016. Οι κύριοι δείκτες είναι ουσιαστικά ένα σύνθετος δείκτης που λέγεται Market Performance Index, δείκτης επιδόσης της αγοράς, έχει αυτέ τι πέντε συνιστώσει που βλέπετε εδώ τη συγκριτιμότητα των προσφαρών, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές στην αγορά, την εμπιστοσύνη στους παρόχους υπηρεσιών, στους λιανέμπορους για να σεβαστούν τους κανόνες προστασίας του καταναλωτή, το βαθμό με τον οποίο οι προσδοκίες τους καλύπτονται στην αντίστοιχη αγορά, το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι καταναλωτές με την επιλογή που έχουν μεταξύ διάφορων παρόχων και ουσιαστικά η ζημία που υφίστανται οι λόγω των ε, προβλημάτων που συναντούν στην αγορά. Έχουμε λοιπόν ένα σύνθετο δίκτυ. Όπως σας είπα, είχαμε μεθοδολογική αναθεώρηση και τα συμπεράσματα ήταν ότι είναι εύρωστος ο δείκτης. Έχουμε όμως εισαγάγει κάποιες βελτιώσεις. Μία από αυτές είναι ότι η σημασία των ε, διάφορων συνιστώσεων και το πώς δίνονται στο συνολικό δίκτυ ε, ουσιαστικά φαίνονται από την ε, ίδια την ανταπόκριση. Το κύριο, το κύριο πόρισμα είναι το εξής. έχουμε συνολική βελτίωση στη λειτουργία των καταναλωτικών αγορών από την καταναλωτική σκοπιά. Και εδώ βλέπουμε επιτάχυνση μιας θετική τάσης που παρατηρήθηκε από το 2010. Επίσης, βλέπουμε ότι οι υπηρεσίες βελτιώνονται ταχύτερα μεταξύ 2013 και 2015 από τη αγορά των αγαθών, όπου μειώνεται το κενό, το χάσμα αυξανόταν σε όλα τα προηγούμενα κύματα. Και αναρωτηθήκαμε τι μπορεί να εξηγήσει αυτή την αύξηση στην επίδοση. Το κύριο συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε είναι, παίρνουμε το σχάρι, εξετάζουμε αν οι βελτιωμένε οικονομικέ συνθήκε και ανάκαμψη από την κρίση μπορεί να το εξηγήσει το φαινόμενο αυτό. Και οι συσχετισμοί που βρήκαμε δεν υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. Συμπεράναμε λοιπόν ότι ίσως οφείλεται εν μέρη στις μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στα κράτη-μέλη. Διαφορετικέ μεταρρυθμίσεις που ουσιαστικά παρουσιάζουν κάποια αποτελέσματα και βελτιώνουν την εμπειρία των καταναλωτών. Βλέπετε εδώ πώς ε, διάφορες ομαδοποιήσεις αγορών έχουν εξελιχθεί και βλέπετε ότι την ταχύτερη αύξηση την είχαν οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όμως ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα ισομεδοποιήσεις έχουμε αυτό που έχει τις χαμηλότερες επιδόσεις. Ποια είναι η κινητήριος δύναμη αυτής της αύξησης. Είναι ιδίως μια αύξηση στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών στους λιανέμπορους, ε, ότι θα σεβαστούν τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και αύξηση του βαθμού στο οποίο καλύπτονται οι προσδοκίες των καταναλωτών και είχαμε και σημαντική αύξηση στη συγκρισιμότητα των διάφορων προσφορών. Βλέπετε λοιπόν εδώ στη διαφάνεια πως ε, το 2015 έχουμε επιτάχυνση των προηγούμενων εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά στο ποιε αγορέ έχουν τις καλύτερε επιδόσεις και ποιε έχουν μεγεθυνθεί περισσότερο. Θα δείτε εδώ τα αποτελέσματα. Έχουμε εδώ τις αγορές που είναι στο top 3, είναι οι διακοπές, οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας, πολιτιστικές ψυχαγωγίες και οι εμπορικές αθλητικές υπηρεσίες, αυτές που έχουν τις χειρότερες είναι οι υποθήκες και τα επενδυτικά προϊόντα. Αυτά τα τρία ε, είναι και οι υπηρεσίε, ε, συγγνώμη, στο, ε, στα κίνητα. Αυτές οι τρεις είναι στη τελευταία κατάταξη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τα αγαθά, τα βιβλία, τα περιοδικά, εφημερίδες, ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι και τα αγαθά ψυχαγωγίας. Επίσης, οι τρεις χειρότερες είναι τα καύσιμα, τα προϊόντα κρέατος και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Βλέπουμε βέβαια ότι η υψηλότερη αύξηση μεταξύ όλων των αγορών σημειώθηκε για τις πιστοτικές κάρτες στα δάνεια και για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και επίσης και υπηρεσίες ε, των τρένων είναι σημαντική αύξηση. Τώρα αν δούμε τις ομάδες αγορών στις ε, ομαδοποιήσεις, σε αυτό το γράφημα βλέπετε πόσο έχει αυξηθεί η επίδοση σε αυτές τις αγορές. Βλέπετε ότι το κλάστερ που λέμε τραπεζικές υπηρεσίες, που είναι ουσιαστικά ε, ένα σύνολο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση έχει σημειώσει αύξηση και στο οριζόντιο επίπεδο βλέπετε ότι παραδείγματο χάρη οι ψυχολογικές υπηρεσίες ε, έχουν αυξηθεί το λιγότερο αλλά έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το κύμα. Βλέπετε εδώ μια διαφορετική εικόνα για την αγορά των αγαθών όπου βλέπουμε ότι τα κλάστερ, ένα από τα κλάστερ που τα πάνε καλύτερα, τα αγαθά τα πάνε καλύτερα και επίσης τα αγαθά στον τομέα της ακτοκινητοβιομηχανίας έχουν αυξηθεί πολύ αλλά δεν έχουν και πολύ καλές επιδόσεις και εδώ μιλάμε για τα νέα αυτοκίνητα και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αλλά και τα καύσιμα. Όσα σας εξήγησα μέχρι τώρα είναι μια συνολική εικόνα όλων των 28 χωρών μερών της Ένωσης, όμως υπάρχουν σημαντικές αποκλήσεις σε ό,τι αφορά την απόδοση διαφόρων αγορών σε διάφορες χώρες. Στην διαφάνεια βλέπετε την εικόνα τρεις αγορές με τις μεγαλύτερες αποκλήσεις σε ό,τι αφορά την απόδοση. Βλέπετε οι πρώτες πέντε χώρες και, η δεύτερη, και στη δεύτερη σειρά οι κάτω πέντε χώρες και η μεγαλύτερη απόκληση, η μεγαλύτερη διαφορά είναι στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 34,1%. Επίσης, μεγάλη, μεγάλες αποκλήσεις στις ε, ε, υπηρεσίες παροχής νερού καθώς και στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος σε ό,τι αφορά την βελτίωση της απόδοσης των αγορών, στα πλαίσια βέβαια πάντα της ενίας αγοράς. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, ανά αγορά, όπως είπα, βελτιώθηκαν περισσότερο από όλες, αλλά παραμένουν σε χαμηλή απόδοση οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η ψηλή εμπιστοσύνη των, ε, μάλλον ε, ζημία των καταναλωτών στις ε, τηλεπικοινωνίες διότι ε, σημειώνονται σημαντικά προβλήματα πολύ συχνά. Εκεί έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών που ε, καταγγέλουν. Άλλα ευρήματα λένε για πρώτη φορά υπηρεσίες μεσητών αν πάτω όπως λέμε, έχουν δηλαδή τη χαμηλότερη απόδοση. Βλέπουμε μια αύξηση για πρώτη φορά όπου οι, ε, σε τομείς όπου οι καταναλωτές αλλάζουν πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος. Για πρώτη φορά μετά το 2010 λοιπόν έχουμε περισσότερους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο, ιδίω όπως είπα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το 2011 λοιπόν πρώτη φορά, σε ασφαλιστικές υπηρεσίες έχουμε την μεγαλύτερη ζημία όταν προκαλούνται προβλήματα, όμως δεν σημειώνονται τόσο συχνά προβλήματα. Όμως, για να σημειωθεί πρόβλημα πρέπει να συμβεί ένα σχετικά ε, απίθανο γεγονός. Ε, μίλησα για αυτό το switching, την αλλαγή δηλαδή παρόχου. 11% το 2015 καταναλωτών, αυξητική τάση σε σχέση με το 2013 αναστρέφει προηγούμενη τάση 2010-2011. Η ψηλότερη, το ψηλότερο ποσοστό switching είναι σε υπηρεσίες αναψυχής και το χαμηλότερο είναι σε τραπεζικές υπηρεσίες. Και κάτω-κάτω είναι οι υποθήκες, όπου μόνο 7% έχουν αλλάξει πάροχο της υπηρεσίας αυτής. Αυτό το switching, ο ίδιος ο ρυθμός switching δεν είναι επαρκής για να εξηγήσει πόσο καλά αποδίδει μια αγορά. Ερωτούμε λοιπόν και άλλες, κάνουμε και άλλες ερωτήσεις σχετικές με την αλλαγή αυτή, με το switching, δηλαδή πόσο εύκολο φάνηκε στον καταναλωτή να κάνει την αλλαγή αυτή και για αυτούς που δεν άλλαξαν, για ποιους λόγους δεν άλλαξαν. Σε ό,τι αφορά την ευκολία του switching, εξετάζουμε τις ομαδοποιήσεις αγορών. Το switching αξιολογείται ως ευκολότερο για υπηρεσίες ασφαλιστικές και ψυχαγωγίας. Και τους χαμηλότερους βαθμούς τους λαμβάνει στις τηλεπικοινωνίες. Γίνεται λοιπόν δυσκολότερα εκεί. Η ανάλυση αναγορά δείχνει ότι οι καταναλωτές βρίσκουν ευκολότερο να αλλάξουν πάροχο στον εμπορικό αθλητισμό για τα οχήματα, ενώ αγορές όπως υποθηκών ε, σταθερής τηλεφωνίας, επενδυτικών προϊόντων, αξιογράφων κλπ. Εκεί είναι δυσκολότερο. Πάλι στο κάτω-κάτω της αγοράς βρίσκεται ο τομέας των υποθηκών. Για πρώτη φορά, σε τούτην εδώ την έκδοση του πίνακος επιδόσεων, έχουμε κάνει και μια πολυμερή αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη και τα κοινωνικά δημογραφικά στοιχεία των καταναλωτών. Στην ανάλυση αυτή, αυτή η ανάλυση μάλλον είναι διαφορετική, με την έννοια ότι επιτρέπει να υπολογιστεί το καθαρό αποτέλεσμα των διαφόρων χαρακτηριστικών με έλεγχο από πλευρά άλλων χαρακτηριστικών. Και αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι ότι η οικονομική κατάσταση είναι και εκείνη η οποία έχει τη μεγαλύτερη σχετική επιρροή στην συνολική απόδοση της αγοράς όπως κρίνεται από την πλευρά των καταναλωτών. οι καταναλωτές που βρίσκουν δηλαδή δύσκολο να τα βγάλουν πέρα, κρίνουν την απόδοση αγοράς λιγότερο ευνοϊκά. Και αυτό ενδέχεται να έχει σχέση με το γεγονός ότι έχουν και περιορισμένη πρόσβαση οι καταναλωτές αυτοί σε ορισμένα είδη αγαθών. Τον Φεβρουάριο φέτος εκδώσαμε και μελέτη για την ε, τροτότητα των καταναλωτών, το ευάλωτο των καταναλωτών, που ε, έρχεται σε επίρρωση των ε, στοιχείων αυτών. Δηλαδή, καταναλωτές που έχουν λιγότερο εισόδημα, έχουν προβλήματα συχνά πρόσβασης, για παράδειγμα τους αρνούνται να τους χορηγήσουν δάνεια, τους αρνούνται να τους εκδώσουν πιστοτικές κάρτες και ούτω καθεξής. Και αυτό ανεβρίσκεται σε όλες τις διαστάσεις του, της ευαλωτότητας. Η παιδεία, η εκπαίδευση δηλαδή, δείχνει επίσης να έχει ε, μια επιρροή στην κρίση της απόδοσης της αγοράς που κάνουν οι καταναλωτές και υπάρχει αρνητικός συσχετισμός μεταξύ των βαθμών που λαμβάνει η απόδοση της αγοράς και της ε, παιδείας και της εκπαίδευσης. Άνθρωποι υψηλότερης παιδείας έχουν μεγαλύτερες ε, προσδοκίες και δίνουν ε, ε, χαμηλότερους βαθμούς. Εξετάζουμε τώρα και άλλους δείκτες που δεν αποτελούν μέρος του Main Composite Index, αλλά δείχνουν πώς ε, διασυνδέονται οι διάφορες ε, συνιστώσεις. Όταν αναλύουμε τις τιμές βλέπουμε για παράδειγμα ότι υπάρχει ένα συσχετισμός μεταξύ της ευκολίας αλλαγής, switching, και του επίπεδου τιμών. Δηλαδή οι τιμές είναι χαμηλότερες σε χώρες όπου η αλλαγή παρόχων υπηρεσιών κρίνεται ως ευκολότερη και σε ορισμένες αγορές όπως ηλεκτρονικών προϊόντων, μεγάλων οικιακών συσκευών, βιβλίων, εφημερίδων, καθώς και ταχυδρομικών υπηρεσιών, καθώς και οχημάτων και ασφαλίσεων, βλέπουμε συσχετισμό μεταξύ του πώς κρίνουν τις υπηρεσίες αυτές οι καταναλωτές και των τιμών. χαμηλότερε τιμέ και μεγαλύτερη ευκολία αλλαγή από πλευρά καταναλωτών. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα ε, στοιχεία σχετικά με, την, με τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών για το 2016. Αυτά τα έχετε και στην ιστοσελίδα μας βεβαίως διαθέσιμα και πολύ ευχαρίστως να απαντήσω σε ενδεχόμενες ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Should I... Θέλετε να προχωρήσει την επομένη ε, παρουσίαση. Ναι, να συνεχίσουμε τη δεύτερη παρουσίαση. Εκτός αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Α, η Εύλην Κέπχαρτ έχει μια ερώτηση. Κοιτάξτε, ερώτηση για τους αριθμούς που μας δώσατε σχετικά με τις αλλαγές των παρόχων. Είπατε ότι στον τομέα των ασφαλίσεων είναι ευκολότερο ή ταχύτερο, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Αυτά βλέπω από τον πίνακά σας. Εξετάσατε επίσης αν υπάρχει συσχετισμός και με τις αλλαγές των συνθήκων διότι των συμβάσεων, συγγνώμη, διότι προσφέρονται με νέες συμβάσεις στις τηλεπικοινωνίες, αλλά Ταυτόχρονα δεν εμπλέκεται η σύμβαση την οποία έχετε από μακρού χρόνου, ενώ στις ασφαλίσεις όταν γίνεται αλλαγή της συμβάσεως δίνει αυτομάτως το δικαίωμα στον καταναλωτή να την καταγγείλει χωρίς να περιμένει την λήξη της. Το εξετάσατε αυτό γιατί αυτό παίζει και ένα ρόλο στην αιτιολόγηση. Γιατί δηλαδή γιατί στον ένα τομέα γίνονται ε, συχνότερες αλλαγές παρόχων από ό,τι σε έναν άλλο. slide... Κοιτάξτε, αυτά που βλέπω εγώ από την ε, διαφάνεια σας αυτή, ε, λέτε ότι είναι ικανοποιημένοι, δηλαδή μετά την ικανοποίηση όλων των καταναλωτών σε όλους τους τομείς, αλλά το τελευταίο που είπατε, συνδέει την ικανοποίηση των καταναλωτών από τη δυνατότητα επιλογών. Και λέτε ότι εκεί όπου οι καταναλωτές έχουν περισσότερες επιλογές, βλέπουν και τις τιμές να μειώνονται και έχουν και υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησεως. Μπορώ με τον τρόπο, από τον απλουστευτικό κάπως αυτόν τον τρόπο, να συνοψίσω τα όσα είπατε με πολλές λεπτομέρειες. Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Πρώτα για το switching. Εδώ υπάρχουν δύο είδη switching. Το ένα είναι το εξωτερικό switching που αλλάζει κανείς τον πάροχο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε και το προϊόν, δηλαδή να παραμείνετε στον ίδιο ε, πάροχο, αλλά με διαφορετική σύμβαση. Internal switching δηλαδή στα αγγλικά. Εδώ εμείς δεν μετρήσαμε το internal switching, εξετάσαμε μόνο στην ε, ε, έρευνα αυτή το εξωτερικό switching. Ωστόσο, για το επόμενο κύμα μελετούμε να εξετάσουμε και το εσωτερικό switching, τον βαθμό δηλαδή όπου άλλαξαν προϊόν που καταναλώνουν οι καταναλωτές με τον ίδιο πάροχο. Και όταν ρωτούμε βέβαια και τους λόγους για τους οποίους δεν άλλαξαν πάροχο, σκεπτόμαστε να βάλουμε και αυτή τη δυνατότητα, ότι δηλαδή ενδεχομένως τους προσφέρθηκε μια βελτιωμένη σύμβαση από την ίδια εταιρεία παροχής υπηρεσιών. Στο παρελθόν, πάντως, κάναμε έρευνα και για το εξωτερικό switching, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες και έχουμε σχετικές εκθέσεις για τους δείκτες αυτούς, αλλά βέβαια συγκρίνουμε μόνο τα όσα είναι δυνατόν να συγκριθούν. Ε, πρέπει να έχουμε κάνει τις ίδιες ερωτήσεις για να μπορούμε δηλαδή να συγκρίνουμε. Όταν μιλούμε λοιπόν για ένα ποσοστό ανθρώπων που άλλαξαν, που έχει αυξηθεί, εννοούμε αυτό το εξωτερικό switching. Δεν μπορούμε βέβαια μόνο από το ποσοστό του switching να αντλήσουμε ε, οριστικά συμπεράσματα. Γι' αυτό εξετάζουμε και την ευκολία ε, switching από αυτούς που προέβησαν στην αλλαγή και τους λόγους για τους οποίους δεν έκαναν την αλλαγή. Όσοι άλλαξαν πάροχο λένε ότι είναι ευκολότερο να αλλάξουν στις διασφαλίσεις παρά στις τηλεπικοινωνίες. Και βεβαίω οι λόγοι που αναφέρατε μπορεί να είναι πράγματι ισχυροί σε ό,τι αφορά δηλαδή το είδος των συμβάσεων. Τώρα, εάν έχει αυξηθεί η ικανοποίηση των καταναλωτών σε όλους τους τομείς, συνολικά ο δείκτης αποδόσεως των αγορών, που δεν είναι μόνο η ικανοποίηση των καταναλωτών, αλλά και συγκεκριμένες εμπειρίες, συγκρισιμότητα, επιλογή, εμπιστοσύνη στους ε, παρόχους, ζημία που υφίσταται ο καταναλωτής όταν σημειώνονται προβλήματα, έχουν αυξηθεί και αυτά σε όλες τις αγορές που εξετάσαμε σε αυτό το κύμα. Σε ορισμένες λιγότερο, σε ορισμένες όμως αρκετά σημαντικά. Πάντως, όταν εξετάζουμε αγορές και χώρες, βρίσκουμε παραδείγματα όπου σε συγκεκριμένες χώρες Κάποιες αγορές είδαν να μειώνονται οι αποδόσεις τους. Η ανάλυση των ε, ε, δεδομένων δηλαδή δείχνουν, ε, δείχνει μια πιο συγκεκριμένη εικόνα και αυτό ισχύει και για την εξέλιξη από, την, από το προηγούμενο κύμαση του σε τούτο εδώ. Σε ό,τι αφορά την επιλογή έχουμε εισαγάγει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο τίθεται η ερώτηση περί επιλογής. Δεν ρωτούμε δηλαδή αναγκαστικά αν υπάρχουν περισσότερες ή λιγότερες επιλογές, αλλά πόσο ικανοποιημένος είναι ο καταναλωτής από την υφισταμένη επιλογή. Διότι σκεπτόμαστε, και αυτό μας το είπαν πολλοί stakeholder, σκεπτόμαστε ότι περισσότερες επιλογές δεν είναι πάντοτε απαραίτητα καλύτερες για τους καταναλωτές. Απαιτούνται και άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, πόσο συγκρίσιμες είναι οι επιλογές, διαφάνεια, εμπιστοσύνη. Το ερώτημα λοιπόν για τις επιλογές ήταν περισσότερο πόσο ικανοποιημένοι είναι οι καταναλωτές από τις υφιστάμενες επιλογές. Και βλέπουμε όντως ότι σε χώρες όπου απαντούν ότι είναι ικανοποιημένοι με τις υφιστάμενες επιλογές σε εκείνες τις συγκεκριμένες αγορές, στις αγορές που σημειώνονται εκεί, αυτό συσχετίζεται και με χαμηλότερες τιμές. Το οποίο είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να ερευνούμε και στις επόμενες φάσεις για να δούμε και πόσο στιβαρή είναι αυτή η συσχετισμή και θα εξετάσουμε και άλλες αγορές βεβαίως τις επόμενες φορές για να δούμε αν και σε άλλες αγορές εμφανίζονται ε, οι ίδιες τάσεις. Επανέρχεται η κυρία Γκέπχαρτ. Ε, πάλι να επαναλάβω μια ερώτηση. Όντω αναφερόμουν και εγώ στις εξωτερικές αλλαγέ external switch δηλαδή, και δεν πρέπει να αναμειγνύει κανεί το εξωτερικό με το εσωτερικό. Αλλά έχω μια ερώτηση ακόμη. Ακούω συχνά περί προστασίας καταναλωτών που σημαίνει χαμηλότερες τιμές. Στην έρευνά σας παίζει ένα ρόλο και η ποιότητα των υπηρεσιών και ε, των ε, προϊόντων ή καθαρά και μόνο το ύψος των τιμών. απάντηση της Επιτροπής. Οι τιμές δεν είναι τμήμα του δίκτυα αποδοτικότητας των αγορών. Πρόσθετος δείκτης που εξετάζουμε μέσα στα πλαίσια ε, του υπολογισμού του δίκτυ. Η ποιότητα. Υπάρχει μάλλον μία ερώτηση η οποία εντάσσεται στον Market Performance Indicator και λέει κατά πόσον η αγορά ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών. Το προηγούμενο το δεκάμινο, πριν από που προηγείται δηλαδή της έρευνας. Αυτή είναι μια από τις συνιστώσεις που έδειξαν σημαντική αύξηση του 2015. Σημαντικός μοχλός δηλαδή, μαζί με την εμπιστοσύνη, η ε, φροντίδα δηλαδή που ε, επιφέρουν οι ε, πάροχοι υπηρεσιών, οι έμποροι κτλ. στις απαιτήσεις των καταναλωτών. Κάνουμε και έρευνες follow-up αγορών που έχουν χαμηλή αποδοτικότητα για να αντιληφθούμε ποιοι είναι οι λόγοι της έλλειψης ικανοποίησης του καταναλωτή. Αυτό ε, μπορώ να σας απαντήσω όσο αφορά την ποιότητα. Δηλαδή, εάν η αγορά ικανοποιεί τις προσδοκίες των καταναλωτών. Αν ανταποκρίνεται τις προσδοκίες των καταναλωτών. Ας περάσουμε στη δεύτερη παρουσία. Αναρωτιέμαι κατά πόσο θα μπορούσε κανείς να μάθει περισσότερα αν εξέτασε τα δεδομένα αναχώρα. Γιατί έχουμε τώρα γενικές δηλώσεις, ενώ θα μας βοηθούσε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν οι καταναλωτές. Εντάξει, όχι τώρα, αλλά πάντως αν θα μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα μαθήματα χρησιμοποιώντας τα δεδομένα αναχώρα, καλό θα ήταν. Δεύτερη παρουσίαση τώρα. Ευχαριστώ. Για αυτό το τελευταίο που είπατε, συμφωνώ μαζί σας. Και στο βαθμολόγιο υπάρχουν φάκελοι αναχώρα, δελτία αναχώρα, με περισσότερες λεπτομέρειες αναχώρα, που δείχνουν τι επιδόσεις έχει αγορά κάθε χρόνο, αναχώρα, σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Και έτσι βλέπουμε αν υπάρχουν αγορές όπου κάποια χώρα έχει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις και αλλού όχι. Είναι μία ανακεφαλαίωση. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ειδικέ ε, αγορές υπάρχουν. Τώρα, η αξιολόγηση των ε, επιπτώσεων ε, του καταναλωτή στην εκπόνηση πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι κάτι που αποφασίσαμε πέρυσι στα πλαίσια του πακέτου για την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αρχίζουμε από το δεδομένο ότι η ποιότητα των πολιτικών επιλογών βελτιώνεται αν τηρήσουμε τις αρχές της καλύτερης νομοθετικής ρύθμισης. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές λοιπόν και οι σχετικές εργαλειοθήκες είναι κάτι που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε οι πολιτικές μας να βασίζονται σε δεδομένα και σε συγκεκριμένες πληροφορίες και να αποφασίζουμε και έγκαιρα γιατί βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν. Οι κύριες κατευθυντήριε γραμμές για την καλύτερη νομοθετική ρύθμιση έχουν ε, υποχρεωτικές ε, δεσμεύσει και εργαλειοθήκες αποτελούν επιπλέον κατευθυντήριε γραμμές και συμβουλές όσον αφορά τη λειτουργία της μεθόδου. Η αξιολόγηση λοιπόν έχει να κάνει και με τα εργαλεία, αν και αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, λέγεται ρητά. Πάντως ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι ότι υπάρχει όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για το εργαλείο αυτό, το Consumer Impact Assessment Tool. Αποτελείται από τρία στοιχεία. Το ένα είναι η λογική της αξιολόγησης αυτής, γιατί χρειάζεται να γίνεται. Έπειτα έχουμε τις διάφορες διαστάσεις, γιατί πρόκειται για κάτι πολυδιάστατο. Και στη συνέχεια έχουμε διαθέσιμες μέθοδοι και εργαλεία για να γίνει η αξιολόγηση αυτή. Πρέπει να αξιολογούμε σωστά τις επιπτώσεις αυτές είναι μια οριζόντια ανησυχία γιατί έχει να κάνει με πολλές και διάφορες πολιτικές. Και είναι αλήθεια κυρίως για προϊόντα και αγορές που γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Επίσης, ηλικιακά μεγαλώνει η κοινωνία μας. Υπάρχουν και οικονομικά ευάλωτοι πληθυσμοί ναι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τις επιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Πρέπει να στηρίξουμε και μεθόδους πιο βιώσιμης κατανάλωσης, την υπερπληροφόρηση, αλλά και τις νέες ανάγκες για να μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές την καλύτερη επιλογή στα πλαίσια μιας ελεύθερης αγοράς. Το εργαλείο τώρα διαρθρώνεται γύρω από τρεις άξονες. Πρώτο, μπορεί να επηρεαστεί η δυνατότητα να υποφεληθεί ο καταναλωτής από την εσωτερική αγορά. Αυτό έχει να κάνει με την άρση των συνόρων. Το key blocking που λέμε ή έχει να κάνει με το που κατοικεί ο καταναλωτής. Έπειτα επηρεάζονται οι τιμές, η ποιότητα, η διαθεσιμότητα, η επιλογή των αγαθών και των υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες μειώνουν το κόστος. Σημαντικό αυτό. Να που είμαστε σε οικονομική κρίση. Και επίσης είναι το θέμα της επιλογής, ελεύθερης επιλογής του καταναλωτή. Μπορεί να επηρεαστεί η εμπιστοσύνη, η γνώση, η προστασία του καταναλωτή. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες μειώνουν την ασυμμετρία στην ενημέρωση ή μειώνουν το κόστος. Ή μπορεί να γίνει διόρθωση στρεβλώσεων στην αγορά. Υπάρχουν αγορές οι οποίες έχουν τέτοια συμμετρία στην πληροφόρηση. Αυτοκινητοβιομηχανία, στεγαστικά, ε, τρόφιμα και άλλα. Εμπιστοσύνη. Προκειμένου να τηρούνται τα δικαιώματα των καταναλωτών και να υπάρχουν και διαδικασίες ε, διόρθωσης εφόσον ε, έχει υπάρξει ζημιά στον καταναλωτή, να μπορεί αυτός να αποζημιωθεί. Πολύ σημαντικό αυτό, τώρα που έχουμε και την ψηφιακή επανάσταση, γιατί έτσι διασυνοριακά μπορεί να ψωνίζει πιο εύκολο ο καταναλωτής, οπότε πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στην διαδικασία αυτή της αγοράς online. Μπορεί να επηρεαστεί η ασφάλεια, η... Εδώ έχουμε να κάνουμε με διάφορα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στην διαφήμιση. Για να μπορούν δηλαδή οι καταναλωτές να συγκρίνουν καλύτερα τα προϊόντα και να τους δίνεται κάποια κατεύθυνση ώστε να κάνουν υπεύθυνα την επιλογή τους διασυνοριακά. Μπορεί να επηρεαστούν οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές. Είναι σημαντικό να δούμε οι ευάλωτοι καταναλωτές πώς επηρεάζονται από μια αλλαγή. Μπορεί να έχει να κάνει και με την υγεία τους και με την οικονομική τους ε, κατάσταση. Το να είναι ευάλωτο ο καταναλωτή σημαίνει ότι μπορεί να ανήκει σε μία είτε ηλικιακή είτε κοινωνικο-οικονομική ομάδα όπου να μην έχει επαρκώς τη δυνατότητα να κάνει ελεύθερες επιλογές. Αλλά είναι και μία δυναμική έννοια, γιατί οποιοδήποτε καταναλωτής κάτω από κάποιες συνθήκες μπορεί να γίνει ένας ευάλωτος καταναλωτής με κάποιες αλλαγές στη ζωή του, ή επειδή ακριβώς είναι τόσο περίπλοκες μερικές φορές οι πρακτικές στην αγορά ή τα προϊόντα με τα οποία ασχολείται. Τώρα, ποιες έννοιες κλειδί χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση. Η... Τα ωφέλη του καταναλωτή από τα αγαθά και τις υπηρεσίες. πόσο μπορεί να αποφεληθεί από αυτά δηλαδή. Έπειτα η ψηφιοποίηση της αγοράς επιτρέπει στον καταναλωτή να αποφεληθεί από ευρύτερη επιλογή προϊόντων και αγαθών, γιατί έχει πρόσβαση σε πιο φτηνές τιμές άμα ψάξει. Η μεγαλύτερη επιλογή τους ε, προσφέρει περισσότερο πλούτο ε, αγαθών η εμπειρία επίσης του καταναλωτή. Τι ζημιά μπορεί να υποστεί τώρα. Μπορεί να υποστεί διαρθρωτική ζημιά που έχει να κάνει με τη γενική λειτουργία της αγοράς ή μπορεί να έχει να κάνει με προβλήματα του ίδιου του καταναλωτή απέναντι στην αγορά. Και τέλος υπάρχουν και οι συνθήκες του καταναλωτή. Περιλαμβάνεται και αυτό στο βαθμολόγιο για να μπορέσει να έχει κατανοητήσει όσο γίνεται περισσότερες επιλογές στις διαστάσεις που είπαμε και την προηγούμενη φορά γνώση, εμπιστοσύνη, συμμόρφωση και τέλος επίλυση διαφορών. Αυτές οι διαστάσεις είναι τα τρία στάδια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ε, συναλλαγή. Προσφέρουμε επίσης και μη λειτουργία helpdesk. Και αυτό είναι ένα ζωντανό έντυπο. Μερικές φορές απαιτεί περισσότερη βοήθεια. Προσφέρουμε λοιπόν βοήθεια, κυρίως όταν πρόκειται για τον εντοπισμό συγκεκριμένων δεδομένων για έρευνες, για πρόσφαση των καταναλωτών αν χρειάζεται διαβούλευση. Ε, μεθοδολογική βοήθεια επίσης όσον αφορά τις μεθόδους και τα εργαλεία. Όσον αφορά τα μεθοδολογικά εργαλεία και οι πηγές δεδομένων, εδώ ένα βαθμολόγιο είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δεδομένα από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση εναρμονισμένα δεδομένα επίσης για τις προσφυγές των ε, καταναλωτών. Καταγράφονται με συγκεκριμένο τρόπο βάσει της σύστασης της Επιτροπής του 2010. Συγκεντρώνουμε λοιπόν τέτοια δεδομένα και τα βάζουμε στην ε, βάση δεδομένων. Εξετάζουμε εναρμονισμένα δεδομένα, όπως είπαμε και τις προσφυγές, έχουμε την ε, βάση δεδομένων RAPEX και γίνονται μελέτες και σε βάθος. Και η τελευταία διαφάνεια. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το roll-out του εργαλείου αυτού. Είμαστε σε επαφές με διάφορες πολιτικές της Επιτροπής και όσον αφορά μέχρι τώρα με την εφαρμογή αυτού του εργαλείου, εμφανίστε στην ανθεώρηση του handbook για την αξιολόγηση. Είναι το χειρίδιο που καθοδηγεί δηλαδή τέτοιες ε, εκθέσεις επιπτώσεων, μελέτες επιπτώσεων για βιωσιμότητα εμπορίου, για παράδειγμα, όπως επίσης εκτίμηση επιπτώσεων για πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν ε, με εμπορική δικαιοσύνη ή θέματα ΦΠΑ. Κάποια παραδείγματα δηλαδή που έχουν χρησιμοποιηθεί αυτά τα εργαλεία και που έχουν ε, φέρει καρπούς. Προσφέρουμε βοήθεια λοιπόν και σε άλλες υπηρεσίες για διάφορες πολιτικές Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά ήταν συναρπαστική η παρουσίαση. Έχω μία ερώτηση σε ό,τι αφορά την ουσιαστική και αναλυτική διαμόρφωση αυτού του consumer welfare της ε, ευημερίας του καταναλωτού. Άκουσα και την ερώτηση της κυρίας Κέπχατ προηγουμένως που της απήντησαν ότι οι οικονομικές πτυχές δεν έπαιξαν ρόλο. Πώς όμως τότε ορίζεται αυτή η ευημερία του καταναλωτού. Θα ήθελα μια διευκρίνηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλετε να επανέλθετε. Η έννοια της ευημερία του καταναλωτή περιγράφεται και στο εργαλείο. Αναφέρεται σε ατομικά φαΐλη που προέρχονται από την κατανάλωση αγαθών υπηρεσιών και τυπικά μετράται μέσω της έννοιας του καταναλωτικού πλεονάσματος που είναι κάτι κοινό οικονομικές μελέτες, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του πόσο ε, ο καταναλωτής προθυμοποιείται να πληρώσει και πόσο πρέπει να πληρώσει για ένα προϊόν. Όταν ε, έχουμε ένα συνολικό μέτρο για τους καταναλωτές, ε, το πλεόνασμα είναι ουσιαστικά ένας δείκτης που μας δείχνει τη συνολική ευημερία του καταναλωτή, έτσι το χρησιμοποιούμε και πρέπει να αναφέρω ότι εις βάθος μελέτες μας για την αγορά προσπαθούν ιδίω ε, να Κάνουν κάποιες εκτιμήσεις σε τομείς όπου μελετάνε τα ωφέλη για τους καταναλωτές από διάφορες παρεμβάσεις στην αγορά ή διάφορα στοιχεία της αγοράς. Βασίζονται επίσης στον ονορισμό του ΣΑ στην ευημερία του καταναλωτή. Δηλαδή χρησιμοποιούμε έννοιες που ισχύουν σήμερα στα οικονομικά. Πρόεδρος, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό το εργαλείο μελέτης αντικτύπου για τους είναι κάτι καινούριο. Κάτι που είναι καλό, γιατί δεν είχαμε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Αλλά ας δούμε την νομοθεσία που εκπονούμε αυτή τη σπονή, που είναι ουσιαστικά η αγορά online ε, των ε, αγαθών, όπου διάφορες χώρες έχουν ε, διάφορα διαφορετικά δίκαια για τον καταναλωτή αυτή τη στιγμή. Κάνατε μία μελέτη αντικτύπου για το φάκελο αυτό και το κάνατε αναχώρα. Γιατί θα θέλαμε να δούμε τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Επίσης, για ποιον ρωτάτε ε, σε ποιον θέτετε τις ερωτήσεις, δηλαδή τους ίδιους τους καταναλωτές ή πρόκειται για ένα ακαδημαϊκό εγχείρημα εντός της Κομισιόν. Είχαμε παραδείγματος χαρή μια διαβούλευση για το refit, για όλο το κεκτημένο, το καταναλωτικό και μόνο 200 από τα 500 εκατομμύρια των καταναλωτών στην Ευρώπη πήραν μέρος στη διαβούλευση και εγώ νομίζω ότι ουσιαστικά μόνο 16 από τις 28 οργανώσεις, μάλλον από τις, οι οργανώσεις 16 από τις 28 χώρες συμμετείχαν. Ποιος απαντά λοιπόν τις ερωτήσεις και ουσιαστικά τι κάνατε σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση που αφορά τα αγαθά και η απάντηση που δόθηκε στον κύριο Σφάπ και η απάντηση που δόθηκε σε μένα είναι κάπως αντιφατικές μεταξύ τους και ίσως κάποια στιγμή θα πρέπει να εμβαθύνουμε. Η δική μου ερώτηση μπαίνει τώρα, αυτή που θα κάνω τώρα δηλαδή, σε μια άλλη κατεύθυνση, ιδίω όσον αφορά την καταναλωτική ευημερία, το consumer welfare. Τι ακριβώς είναι και πώς ορίζεται. Υπάρχει άραγε τρόπος πραγματικά να ε, γίνει ένας ευρωπαϊκός ορισμός αυτής της ευημερίας του καταναλωτού. Ε, βλέπουμε για παράδειγμα ότι το δίκαιο των καταναλωτών διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα. Αυτό δεν είναι ένα σημάδι ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών ανά χώρα μέλος αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Ίσως και η δυνατότητα επιβολής τους των δικαιωμάτων δηλαδή. Βλέπω για παράδειγμα ότι στην Μεγάλη Βρετανία είναι πολύ σημαντικό όταν διαπιστώνονται κάποια λατώματα σε αγαθά, να έχει τη δυνατότητα επιλογής ο καταναλωτής να επιστρέψει το προϊόν ή να λάβει μια χρηματική αποζημίωση. Ενώ στη Γερμανία δεν συζητεί το θέμα, ο έμπορος αποφασίζει ε, ποια επιλογή θέλει να ισχύσει. Άρα πρόκειται λοιπόν για διαφορετική αντιμετώπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ανά χώρα μέλος. Τέτοιες διαφορές πώς είναι δυνατόν να μετρηθούν και να ενταχθούν μέσα σε αυτό το consumer welfare. Εν πάση περιπτώσει πώς αντιμετωπίζετε τέτοια θέματα. Θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας για την ε, πρόταση για την επιγραμμική αγορά υλικών αγαθών. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Έχουμε ουσιαστικά κάνει εις βάθος μελέτες αξιολόγησης του αντικτύπου και έχουμε και ένα μικροοικονομικό μοντέλο που ουσιαστικά εξετάζει τον αντίκτυπο στην οικονομία συνολικά και στην ευημερία των καταναλωτών στις καταναλωτικές τιμές. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι διαθέσιμα και κατανέμονται ανά χώρα και τα διαιρούμε ένα χώρα και έχουμε, ενημερώσει, έχουμε μια ενημερωμένη μελέτη αντικτύπου και υπάρχει και ένα ειδικό παράρτημα της μελέτης αντικτύπου με την ανάλυση αυτή. Τώρα, να αποσαφηνίσω ότι αυτό το εργαλείο που έχουμε αναπτύξει για τη μελέτη αντικτύπου σκοπεύει στοχεύει κυρίως ε, στους άλλους συναδέλφους από την Κομισιόν, από τις άλλες ε, γενικές διευθύνσεις που ίσως να μην ε, γνωρίζουν τόσο καλά την ανάγκη να αξιολογήσουν τις μελέτες αντικτύπου και δεν μπορούν να μην έχουν πλήρη γνώση των μεθόδων. Έτσι λοιπόν, οι άλλες υπηρεσίες είναι η κυρία ομάδα στόχος μας και τώρα προβαίνουμε σε ευαισθητοποίηση και υποστηρίζουμε τη χρήση αυτού του εργαλείου. Ενώ για τις ε, πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η δική μας υπηρεσία Ήδη κάναμε αυτή την ανάλυση στο παρελθόν και χρησιμοποιούμε τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουμε για τους καταναλωτές. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δημόσια διαβούλευση για το refit. Η δημόσια διαβούλευση διαφέρει από μια έρευνα ή από μια έρευνα που βασίζεται κάποιο δείγμα. Έτσι λοιπόν δημόσια διαβούλευση βασικά λαμβάνει κάποιες συνεισφορές από επιλεγμένους ανθρώπους που απαντούν και παίρνουν το χρόνο να κάνουν αυτή τη συνεισφορά, συνήθω πρόκειται για ενδιαφερόμενα μέρη, λιγότερο για μεμονωμένου καταναλωτέ, γιατί ξέρετε το να απαντήσει κάποιο σε μια δημόσια διαβούλευση απαιτεί και ένα επίπεδο εμπειρογνωμοσύνη, γνώση, εξοικείωση με την νομοθεσία. Και πολλοί μεμονωμένοι καταναλωτέ δεν τα διαθέτουν αυτά. Διαφέρει λοιπόν η τεχνική. Και οι ποσότητες είναι μικρότερες από ότι η ποιότητα και η ουσιαστική, το ουσιαστικό input. Γιατί ουσιαστικά εδώ παίρνουμε κάποια στοιχεία βάσει των εμπειριών. Ενώ στις έρευνες που κάνουμε, στις δημοσκοπήσεις και σε άλλα είδη συλλογή δεδομένων, γιατί χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων Μπορεί να αφορούν τις τιμές, μπορεί να αφορούν το είδος των αγορών, κάποια μοντέλα συμπεριφοράς κτλ. Διαβουλεύσεις. Ουσιαστικά κάθε ένα από αυτά τα μέσα έχει τις ιδιαιτερότητές του αλλά δεν θα έλεγα να θεωρήσετε τη δημόσια διαβούλευση ένα είδος έρευνας και ουσιαστικά να πείτε ότι δεν απαντούν πολλοί. Οπομένως, είναι ένα διαφορετικό είδος εγχειρήματο και σε ό,τι αφορά τώρα τι κύριε ερωτήσει, αυτές βασικά θέλουν να προσανατολίσουν την ανάλυση και κάθε ερώτηση, σε κάθε ερώτηση κλειδί δίνουμε μεθόδους και πηγές δεδομένων στο εργαλείο και υποστήριξη για το πώς θα μπορούσε να γίνει η ανάλυση αυτή. Βέβαια, ε, ουσιαστικά η εφαρμογή αυτή έχει να κάνει με ένα checklist που πρέπει να εφαρμόζεται σε μεμενωμένες πολιτικές ανάλογα με τη σκοπιμότητα. σε σχέση με την ερώτηση για την ευημερία των καταναλωτών. Εάν είναι δυνατό να έχουμε έναν ορισμό που να λειτουργεί σε όλα τα κρατη και σε όλους τους πολιτισμούς. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Και ακριβώς ε, ο τρόπος που ορίζεται περιέχει αυτή την ποικιλομορφία. Γιατί το κέρδος της ευημερίας ε, σχετίζεται με το πλεόνασμα. Και τι σημαίνει καταναλωτικό πλεόνασμα. Είναι η διαφορά μεταξύ του τι εγώ θα ήθελα να πληρώσω για ένα προϊόν ή για μια υπηρεσία ως καταναλωτής και ποια είναι η τιμή της αγοράς. Επομένως, η προθυμία του να πληρώσει κανείς, το, το ποσό που θα πληρώσει κανείς, διαφέρει από άτομο σε άτομο. Παραδείγματο χάρη ένα άτομο που θεωρεί ότι αξίζει αυτό το προϊόν μπορεί να πληρώσει την τιμή στην αγορά, αλλά θα έχει ένα μεγαλύτερο πλεόνασμα από ότι ένα άλλο άτομο που υποκειμενικά, υποκειμενικά αποδίδει μικρότερη αξία σε αυτό το προϊόν. Όταν ε, όλα αυτά τα ομαδοποιούμε, μιλάμε για ένα πλεόνασμα καταναλωτή και την ευημερία του καταναλωτή συνολικά. Υπάρχουν ε, διακυμάνσεις, παραδείγματος χάρη, τα κέρδη για τον καταναλωτή θα ήταν να αυξήσουμε το πλεόνασμα του καταναλωτή μέσω παρέμβασης σε διάφορες πολιτικές. Έχουμε μια αρχική κατάσταση και μπορεί να έχουμε μια παρέμβαση πολιτικής που να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές και να αυξήσει την ευημερία των καταναλωτών, αυξάνοντας το πλεόνασμα του καταναλωτή. Βέβαια, θεωρούμε ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, αλλά όπως και να έχει, οι μικρότερες τιμές αυτούς ωφελούν. Ευχαριστούμε. Θα ολοκληρώσω τώρα εδώ τη συνεδρία σας. Ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας και θα ξεκινήσουμε με τους συντονιστές σας. Ευχαριστώ.